Καλώ Καλώς ήρθατε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Ας εγκρίνουμε την ημέρησια διάταξη. Πριν να καλωσορίσω τον πρόεδρο κύριο Ντράγκη, έχω το σύντομες ανακοινώσεις για τις συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις που άρχισαν στην 5η Ιουλίου οι τριμερείς διάλογοι για το CRD5 και CRR2 και CRD5 με διάκριση ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες αντικειμένων πολιτικών, καθαρά τεχνικών και τεχνικοπολιτικών και ούτω καθεξής και στην βάση αυτή χορηγήσαμε εντολή στο τεχνικό επίπεδο για το επόμενο χρονοδιάγραμμα τριμερούς διαλόγου για τις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Και επίσης είχαμε και τον πρώτο τριμερή διάλογο Εμίρ Ρεφίτ στις 4 Ιουλίου που κινήθηκε πολύ θετικά και μας επέτρεψε να συζητήσουμε θέματα συνταξιοδοτικών συστημάτων και έγινε και μια προκατακτική συζήτηση για υποχρεώσει συμψηφισμού. Αυτά θα συνεχιστούν. Τώρα, θα ήθελα να απευθύνω το θερμό καλώ ορίσατε στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριο Μάριο Ντράγκη, για τον δεύτερο νομισματικό διάλογο του έτου. Και βέβαια, διάλογο που ακολουθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Έκτου, όπου ως γνωρίζετε παραμένει αναλύωτο το επιτόκιο στα παρόντα επίπεδα της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2019 και οι καθαρές αγορές του APP που θα έτρεχαν μέχρι τον Σεπτέμβριο για 30 δισεκατομμύρια τον μήνα συνεχίζονται μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 στο επίπεδο των 15 δισεκατομμυρίων. Θα απευθύνω το καλώς ορίσατε και μάλλον καλωσορίζω και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διατήρηση υψηλού επίπεδου Monetary Accommodation και όσοι γνωρίζετε ενώ το πρόγραμμα θα καταργηθεί σταδιακά θα συνεχιστεί με βασικές πληρωμές για μια εκτεταμένη περίοδο, χρονική περίοδο, και θέλω να συγχαρώ επίσης για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε και ανακοινώθηκε στις αγορές η απόφαση αυτή που νομίζω ότι κατενόησαν καλά και αντέδρασαν καλά στην σημαντική αυτή απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τώρα, όπως είπατε και στη συνέντευξη τύπου, ότι έχουμε καθορίσει η ημερομηνία για το APP. Έχουμε τώρα ένα, ε, μια ευρύτερη εργαλειοθήκη εργαλείων για την νομισματική πολιτική μας που ευθυγραμμίζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις υπόλοιπους μεγάλους πιστοτικούς οργανισμούς του κόσμου. Και αυτό είναι ένα σημάδι ανθεκτικότητας της νομισματικής μας ένωσης. Ως γνωρίζει ο πρόεδρος Δράγκη, οι συντονιστές έχουν επιλέξει δύο πρόσθετα θέματα, δηλαδή τις προκλήσεις για την νομισματική πολιτική και τους ε, περιορισμούς της εγγύησης και άλλα στάνταρτ μέτρα. Έχουμε κάνει κάποια προπαρασκευαστική εργασία με συμμετοχή της ομάδας εμπειρογνωμόνων μας. Θα παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα των μελετών μας και να δώσω τώρα το λόγο σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά που είμαι ξανά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής σας. Από την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως υπενθύμησε και ο Πρόεδρος προλίγου, έλαβε σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την επαναστάθμιση της νομισματικής πολιτικής και της σχετικής τάσης μας μετά από το Σεπτέμβριο ενεστώτος έτους. Στα σχόλιά μου σήμερα θα περιγράψω αυτές τις αποφάσεις και θα εξηγήσω την αξιολόγηση του παρόντος οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου, επί του οποίου βασιστήκαμε. Μετά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωζώνη, δράτω με τη ευκαιρία επίση για να συζητήσω το μέλλον τη Οικονομική και Νομισματική μα Ένωση, κατευθυνόμενο προ προτεραιότητε βραχυπρόθεσμε, όπω τα βλέπει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξήθηκε κατά 0,4% η οικονομία της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2018 και αυτό σημειώνει πέντε χρόνια συνεχούς ε, οικονομικής ανάπτυξης. Παραμένουν εστέρες οικονομικές βάσεις. Βέβαια, έχει κάποιος μετριαστεί η ανάπτυξη αρχές του έτους. Η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί αξιοσημείωτα τα τελευταία χρόνια. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 8,4 εκατομμύρια από τα μέσα του 2013 και αναπτύσσεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε στο 8,4% το μήνα Μάιο, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβρη του 2008 και το εργατικό δυναμικό συμμετέχει ε, σε ύψιστο βαθμό στις προσπάθειες. Τώρα προσβλέποντας το μέλλον, η πρόσφατη μακροοικονομική προβολή του ευρωσυστήματος προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη του 2,1% το 2018, 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Υπάρχουν αβεβαιότητες που σχετίζονται με παγκόσμιους παράγοντες συμπεριλαμβανομένες και της απειλής του αυξανόμενου προστατευτισμού και όλα αυτά όλο και ενισχύονται, ο κίνδυνος που περιβάλλει την Ευρωζώνη και τις προβλέψει την Ευρωζώνη παραμένει α, κάπως ισορροπημένη. Βέβαια παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις αρχιπρόθεσμες του Ευρωστάτ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε το 2, κατά 2% τον Ιούνιο από 1,9% τον Μάιο και αυτό ε, δείχνει ότι έχουμε υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Ε, αν εξαιρέσουμε αυτά τα κειμενόμενα προϊόντα, ε, ο πληθωρισμός μειώθηκε από 1,1% το Μαΐο στο 1% τον Ιούνιο. Συνεχιζομένη στις αυξήσεις της ε, αναπτύξης οικονομίας και της απορροφήσεως της χαλάρωσης, βλέπουμε ότι η υποβόσκον πληθωρισμός θα αυξηθεί. Οι πρόσφατες συμφωνίες μισθολογικές στις χώρες δείχνουν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι θετικές δυναμικές. Θα συζητήσω τι προβλέψει του πληθωρισμού λεπτομερέστερα, εξηγώντα την νομισματική πολιτική τη σχετική αποφάση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Τώρα, στην τελευταία συνάντησή μα για την νομισματική πολιτική, το Διοικητικό Αυτό ανέλαβε να κάνει μια επισκόπηση προσεκτική τη μέχρι τούδε επιτευχή σα πρόοδου για την προσαρμογή στον πληθωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε τι εξελίξει των φατοπληθωρισμών εν συγκρίση με, τους, με τα τρία βασικά κριτήρια για τι αγορέ αξιογράφων στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή σύγκληση, εμπιστοσύνη και αντοχή. Όσον αφορά την σύγκληση, οι, προ... οι προβολές του Eurosystem του 2018 του Ιουνίου είδαν ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 1,7% σε κάθε μία από τις επόμενες τριετίες. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά σε προβλέψεις που προβλέπουν ότι θα συγκλίνει ο πληθωρισμός στο στόχο του πληθωρισμού που θα είναι κάτω αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Η υπεποίθησή μας όσον αφορά τη διαδρομή του πληθωρισμού επίσης αυξάνεται. Πρώτα απ' όλα το φάσμα της αβεβαιότητας που περιτριγίζει τις προβολές για τον πληθωρισμό έχει μειωθεί. Δεύτερον, υποβόσκων πληθωρισμός έχει αυξηθεί από πολύ χαμηλά επίπεδα που επικρατούσαν το 2016 και προβλέπεται να αυξηθεί ενώ συνεχίζεται να αυξάνεται, να βελτιώνεται η οικονομία, ενισχύεται η χρήση του δυναμικού και οι αγορές ε, εργασίας ε, γίνονται και πιο, ε, περιορίζονται περισσότερο. Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, ε, η προβολή όσον αφορά την εξέλιξη του πληθωρισμού δείχνουν ότι έχει σταθερή πορεία. Δηλαδή θα αντέξει όσον αφορά μια σταδιακή ε, μείωση της αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Βάσει αυτής της αξιολογήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπέρανε ότι πρόεδρος προς μια βιώσιμη προσαρμογή υπήρξε ουσιαστική μέχρι τούδε και θα πρέπει να συνεχιστεί στην επόμενη περίοδο παρόλο που επιμένουν και απομένουν κάποιες αβεβαιότητες. Γι' αυτό προβλέπουμε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα μειώσουμε τη μία αγορά ε, στοιχείων ενεργητικού από 30 δις στα 15 δις και θα σταματήσουμε την αγορά στοιχείων ενεργητικού το τέλος του Δεκεμβρίου. Αυτό βέβαια με την επιφύλαξη νεωτέρων στοιχείων που θα επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του πληθωρισμού. Το προσδεκόμενο τέλος των αγορών στοιχείων ενεργητικού το Δεκέμβριο του 2018 δεν σημαίνει ότι η νομισματική μας πολιτική πάβει να είναι επεκτατική. Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να συνοδεύει την οικονομική επέκταση και αύξηση και ανάπτυξη για κάποια χρονική περίοδο. Γι' αυτό επιβεβαιώσαμε εκ νέου την επανεπενδυτική μας πολιτική και αυξήσαμε τους προσανατολισμού μας όσον αφορά τα βασικά επιτόκια. Πιο συγκεκριμένα, προτιθέμεθα να διατηρήσουμε την πολιτική μας επανεπενδύσεων των βασικών πληρωμών από οριμάζους αξιόγραφα που αγοράστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγοράς αξιογράφων μια εκτεταμένη περίοδο χρόνου μετά το τέλος της, των αγορών μας στοιχείων ενεργητικού και εν πάση περιπτώσει το βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να διατηρηθούν ε, θετικές συνθήκες ρευστότητας και να έχουμε έναν ευρύ βαθμό νομισματικών ελιγμών και αναμένουμε ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ να παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα τουλάχιστον ε, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2019 και εν πάση περιπτώσει για όσο αυτό χρειαστεί ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διακύμανση του πληθωρισμού θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη με τις τρέχουσες προσδοκίες μιας βιώσιμης πορείας προσαρμογής. Τώρα να στραφώ στο θέμα της διακυβερνήσεως της οικονομικής και νομισματικής ενώσεως. Σε μια εποχή μεγάλης παγκόσμιας αβεβαιότητας είναι πιο σημαντικό τώρα παραποτέ η Ευρώπη να σταθεί ενωμένη. Οι προσπάθειες που έχουμε καταβάλει τα πρόσφατα έτη για να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενώσεως ήδη έχουν καταστήσει την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση πια θεκτική σε κλειδονισμούς. Όμως η Νομισματική μας Ένωση εξακολουθεί να είναι ατελής και παραμένει ευάλωτη. Για να υποστηρίξουμε την εμπιστοσύνη και να συνεχίσουμε την οικονομική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περαιτέρω σύγκληση και ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Πέρασαν σχεδόν ακριβώς μάλλον έξι χρόνια από όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ξεκινήσουν την Τραπεζική Ένωση. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου και έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των κινδύνων και συνεπώς σε, μια, σε ένα πιο σταθερό ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αλλά η Τραπεζική Ένωση δεν είναι ακόμα πλήρης. Η ταχεία προσαρμογή της δέσμης της εκθέσεως για το δέσμι μέτρων για τις τράπεζες ε, χρειάζεται μια ταχεία πορεία τριμερών διαλόγων. Μάλλον καλωσορίζουμε την έγκριση της εκθέσεως για τραπεζικό πακέτο που καλεί για μια ταχεία διαδικασία τριμερούς διαλόγου, διορθώνει ο μιλητής. Η συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που είναι η βάση για το ενιαίο ταμείο για ρευστοποίηση είναι εξίσου σημαντικό και θα δώσει ένα περαιτέρω επίπεδο ασφαλείας για τράπεζε υποεκαθάριση και η θα μπορεί να γίνει αποτελεσματικά χωρί να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όλα αυτά εν σειρά θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τομέα στο, τομέα στο σύνολό του και θα τον σταθεροποιήσουν. Αυτό το μέτρο σταθεροποίηση θα πρέπει να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν και θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχείε διαδικασίε λήψεω αποφάσεων. Σε επικείμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων και των συζητήσεων για ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό εγγύσεω ε, καταθέσεων, να, δεν θα πρέπει να, να μην μα συγκρατήσει η διάκριση μεταξύ τη μείωση του κινδύνου και του επιμερισμού του κινδύνου για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, ουσιαστική μείωση των κινδύνων ήδη έχει λάβει χώρα το επίπεδο 1 ε, των κοινών στοιχείων ενεργητικού σημαντικών τραπεζών που δείχνει την υγεία των τραπεζών είναι 67% υψηλότερος από ό,τι ήταν 100 παρελθόν, εδώ και 10 χρόνια. Περαιτέρω μείωση των κινδύνων έχει δρομολογηθεί με τη μείωση ε, των κόκκινων δανείων και των τοξικών στοιχείων ενεργητικού σε κάποια χαρτοφυλάκια μεγάλων τραπεζών. Δεύτερον, ο επιμερισμό του κινδύνου βοηθά κατά πολύ τη μείωση των κινδύνων. Κοιτάξτε τι γίνεται με την εταιρεία για την ασφάλιση των καταθέσεων των ΗΠΑ, Ομοσπονδιακό Φορέα. Έχει επιλύσει τα προβλήματα 500 τραπεζών χωρίς να δημιουργήσει χρηματοπιστωτική αστάθεια κατά τη διάρκεια της κρίσης και διότι ε, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αντίστοιχος αριθμός για την Ευρωζώνη ήταν 10 φορές χαμηλότερος, που είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο η Ευρωζώνη και ο τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαθροτικά προβλήματα και προκλήσεις. Με άλλα λόγια, εάν ο επιμερισμός του κινδύνου οδηγούσε σε μια τακτική διαχείριση των συνεπιών για την οικονομική σταθερότητα που απορρέουν από τη μείωση του κινδύνου, η μείωση του κινδύνου αυτή καθ' αυτή θα οδηγούσε σε θα κινείται σε πολύ ταχύτερο ρυθμό. Έτσι δε περαιτέρω, ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό εγγύηση καταθέσεων θα απέφευγε τον κίνδυνο αποσταθεροποίησεω ε, λόγω διαφόρων ε, προφητιών που έχουν γίνει σε προηγούμενε περιόδου. Θα μειωνόταν επίση και ο κίνδυνο χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού και έτσι θα υποστήριζε την αποτελεσματικότητα τη νομισματική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμβάλλοντα στην οικονομική σταθερότητα. Με το σωστό πλαίσιο πολιτική, ο επιμερισμό των κινδύνων και η μείωση των κινδύνων ε, ενισχύονται αμοιβαίω. Μια πιο ανθεκτική οικονομική και νομισματική ένωση επίσης θα ωφεληθεί από ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαχειρίσεως των κινδύνων η δέσμευση να ισχυθεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα που ανελήφθη στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφή του Ευρώ είναι κάτι άκρο ευπρόσδεκτο. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια αύξηση τη αποτελεσματικότητα αυτού και ευελιξία αυτού όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τα διατηθέμενα μέσα, σεβόμενο πλήρω τι εντολέ που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να απορροφηθούν οι κλειδονισμοί και να αποφύγουμε μια πλήρη έκρηξη κρίσεω, η Ευρωζώνη θα αφελείται από ε, μια κοινή λειτουργία σταθεροποίηση. Ένα τέτοιο εργαλείο μπορούσε να παράσχει μακροοικονομική υποστήριξη σε περίπτωση ύφεση σε όλη την Ευρωζώνη, διαφυλάσσοντα τη σύγκληση, υποστηρίζοντα ε, σταθεροποιητικέ εθνικέ πολιτικέ και επιτρέποντα τη νομισματική πολιτική να λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, αυτό το μέσο δεν θα έπρεπε να υπονομεύει κίνητρα για τα κράτη-μέλη, ώστε να επιδιώκουν μια ορθή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική και γι' αυτό καλωσορίζουμε θερμά την ανανομένη όθηση που δίνεται σε αυτή τη συζήτηση. Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την Ένωση των, της Αγοράς Κεφαλαίων μπορεί να στηρίξει και τις προτεραιότητες που σας περιέγραψα. Καταρχάς, η Ένωση των Κεφαλαγορών θα ενίσχυε τον επιμερισμό των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ε, αποσβαίνοντας τοπικούς κλειδονισμούς, μειώνοντας την ανάγκη να χρησιμοποιούνται εργαλεία δημόσια σταθεροποίησεως. Δεύτερον, ένα συνεπές πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για βαθιά και ανθεκτική χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Παραδείγματο χάρη, εναρμόνιση και βελτίωση ε, διαφόρων πλαισίων περί αξιοπιστίας και φερεγγιότητας θα μπορούσε να διευκολύνει τις τράπεζες να μετωπίσουν στοιχεία ενεργητικού που δεν αποδίδουν ή που αποδίδουν και θα είναι υποφελής οι τράπεζες. Μια πραγματική κεφαλαγορά, ενωμένη κεφαλαγορά θα μπορούσε να υποστηρίξει βαθύτερη ε, ολοκλήρωση και θα σταθεροποιήσει τις κεφαλαγορές και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε όλου. Πρέπει να τονίσω ότι κανένα από τα αναφερθέντα μέτρα είναι εφικτά αν μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό απαιτεί το ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα παίξουν το ρόλο τους αυξάνοντας την αντοχή των οικονομιών τους και εξυγχρονίζοντας τις οικονομικές τους δομές. Λοιπόν, κλείνοντας, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής υπήρξαν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Εκτιμούμε ότι τα μέτρα τα οποία λάβαμε από τα μέσα του 2014 θα έχουν ένα σωρευτικό αντίκτυπο περίπου 1,9% και στην πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και τον πληθωρισμό για την περίοδο 2016-2020. Τα μέτρα μας διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο ούτω ώστε να φέρουμε τον πληθωρισμό πίσω στη σωστή πορεία σε επίπεδο που είναι κάτω και κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Όμως πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, επίμονοι και συνετή στις πολιτικές μας για να εξασφαλίσουμε το ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε ένα μονοπάτι σταθερό προσαρμογής. Όπως προαναφέρθηκε, διάφοροι κίνδυνοι που ελοχεύουν σχετίζονται με τον κίνδυνο του αυξανόμενου προστατευτισμού. Μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να δρέψει τους καρπούς της οικονομικά ανοιχτής προσεγγίσεως προστατεύοντας τους πολίτες της κατά ανεξέλεγκτου ε, παγκοσμιοποίησεως. Ηγουμένη παραδείγματος η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει ε, την πολυμερή προσπάθεια και το παγκόσμιο εμπόριο που ήταν ακρογωνία η λύθη ε, της αναπτυσσόμενης οικονομικής ευμαρίας τις ε, τελευταίες 7 δεκαετίες. Αλλά για να είμαστε επιτυχείς εξωτερικά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς και ορθή οικονομική διακυβέρνηση εντός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Τράγκη. και για το γεγονός ότι χαιρετήσετε την έγκριση της δέσμης μέτρων για την Τραπεζική Ένωση ε, και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι η ΕΚΤ ε, ε, γνωρίζει ότι υπάρχει συνήθις νομική διαδικασία, υπάρχει ε, κείμενο από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία είναι ισότιμα και θα τους το υπενθυμίσουμε αυτή την εβδομάδα όταν θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Ε, θα τον ε, διεξάγει ο εισηγητής, ο κύριος Χόκμαρ, ο οποίος είναι και ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τα όσα είπατε και για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να συμφωνήσω με μεγάλο τμήμα των όσων είπατε για την ανάγκη για μια ισχυρή τραπεζική ένωση, κεφαλαγορές. Ε, έχω όμως μία ερώτηση ε, πιο ειδική και μία πιο συγκεκριμένη. Η πρώτη ερώτηση αφορά την ανάπτυξη των ε, δανείων τα οποία εξυπηρετούνται και όσον αφορά την προοπτική της αυξημένης σταθερότητας Πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν αυτά τα δάνεια τις ε, γραμμές που θα έπρεπε να είχαν ακολουθήσει. Αν όχι, ποιος νομίζετε ότι είναι ο βασικός λόγος. Το πιο γενικό θέμα είναι βεβαίως ο πληθωρισμός και η μοναδική επεκτατική νομισματική πολιτική που είδαμε εδώ και αρκετό χρόνο. Ξεκίνησε στα εν μέσω βαθέας κρίσεως 2008-2009 ε, και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο τα πρώτα χρόνια της ανάκαμψης. Ε, μετά παρέμεινε στη διάρκεια της ανάκαμψης ε, και όταν η οικονομία άρχισε να βελτιώνεται ε, παρέμεινε και πάλι και όπως βλέπετε έχουμε φτάσει, ε, είπατε κι εσείς, στα υψηλότερα επίπεδα και εξακολουθούμε να έχουμε μια μοναδική, κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε και ακραία επεκτατική νομισματική πολιτική. Η ερώτησή μου είναι έχει νόημα να ακολουθούμε το κριτήριο του πληθωρισμού με τον τρόπο που το ακολουθούμε. Δεν πιστεύετε ότι οι κίνδυνοι γίνονται όλο ένα και μεγαλύτεροι εάν ακολουθούμε αυτή τη μοναδική νομισματική πολιτική εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα και σε χαλεπούς καιρούς και σε καλούς καιρούς. Και τι θα κάνουμε, τι θα κάνετε εσείς όταν τα πράγματα ε, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους έχουμε αυτή την αίσθηση. Αναφερθήκατε στον προστατευτισμό, αλλά και σε έναν ε, αριθμό διαφορετικών ε, βαθμών αβεβαιότητας που έχουμε σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ε, θα ασχοληθείτε με τις συνέπειες αυτές της μοναδικής νομισματικής επεκτατικής πολιτικής, η οποία διατηρείται εδώ και τόσο καιρό και τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε όταν τελικά οι εξελίξεις δεν είναι τόσο καλές όσο θα είναι σήμερα και επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, πιστεύουμε ότι αυτά τα δάνεια θα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατάσταση έχει ε, βελτιωθεί σημαντικά, αλλά φυσικά δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας. Υπάρχουν μια σειρά από υφέρποντες ε, λόγους ε, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ένα από αυτά ήταν ε, η, η ίδια η ύφεση. Αν συνεχιστεί, σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πολλές χώρες. Όχι σε όλες βεβαίως, αλλά σε πολλές χώρες όπου η αύξησή τους επεκτάθηκε λόγω της μεγάλης ύφεσης θα μειωθούν ουσιαστικά αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη συνέχεια. Και φυσικά υπάρχει πληθώρα λόγων. Καταρχά, οι πελάτε ε, τη τράπεζα, ε, ε, η αξιολόγηση των μετοχών στι αγορέ έχει βελτιωθεί, επομένω υπάρχει δυνατότητα για πώληση αυτών των δανείων. Και ο δεύτερο λόγο είναι η εποπτεία. Έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση και ενίσχυση της εποπτείας για τα ε, μη εξυπηρετούμενα, εγώ θα τα αποκαλέσω ότι μη εξυπηρετούμενη έκθεση, δεν είναι μόνο δάνεια και η διαδικασία εξομάλυνσης μας έχει επιτρέψει να αναβαθμίσουμε τις πρακτικές μας και να είναι πιο αποτιτικές. Η πληροφορία, ο διαμόρφωση λοιπόν των νέων αυτών δανείων που θα είναι μη εξυπηρετούμενα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αυξηθεί από ό,τι στο παρελθόν. Το τρίτο θέμα όμως είναι το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες να ε, ξεφορτωθούν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν θέλετε. Και φυσικά υπάρχουν πληθώρα κανόνων και νομοθεσία την οποία θα πρέπει να εγκρίνουμε, να προσαρμοστεί και εξαρτάται φυσικά από την κατάσταση της κάθε χώρας. Αλλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση στην οποία η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε μία εξυπηρετούμενα δάνεια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και ο λόγος είναι ότι η νομοθεσία αυτή τη στιγμή δίνει κίνητρα για την παραμονή αυτών των δανείων, αντί να δίνει κίνητρα για την πώλησή τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τα τρία συστατικά στοιχεία για να υπάρξει μείωση. Αλλά τη διαπιστώνουμε αυτή τη μείωση σε αυτά τα κόκκινα δάνεια και ό,τι βλέπουμε είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό η δεύτερη ερώτηση για τους κινδύνους ε, της ε, νομισματικής μας πολιτικής. Η νομισματική μας πολιτική καταρχάς δεν είναι μοναδική. Είναι η ίδια νομισματική πολιτική που χρησιμοποίησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι εμείς και ε, στην Αγγλία και στην Ιαπωνία δε. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις, ε, τον πιθανό κίνδυνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που μπορεί να προκύψει από την παρατεταμένη των πολύ ε, πολιτική των πολύ χαμηλών επιτοκίων και της ε, ευρύτατης ρευστότητας. Και τα παρακολουθούσαμε αυτά πάρα πολύ προσεκτικά. Προς το παρόν δεν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι σε αυτό το μέτωπο. και παρεμπιπτόντως στους τομείς στους οποίους διαβλέπουμε κάποιους κινδύνους, η απάντησή μας δεν θα ήταν ε, αλλαγή εκβάθρων της νομισματικής πολιτικής, αλλά ε, ε, χρησιμοποίηση των κατάλληλων μακροοικονομικών εργαλείων. Ευχαριστώ, Υπερβάνης Περές. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, Συγγνώμη, τελικά δεν ξέρω, λέει η κυρία Περέ. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση για την ε, διακυβέρνηση της ε, ΕΚΤ και των ε, κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών. Τον Απρίλιο αναφερθήκατε στο δικαστήριο για την περίπτωση του κυβερνήτη της Τράπεζας της Λετωνίας, ο οποίος ε, επάφθηκε ε, για κατάχρηση. Θα ήθελα να ξέρω καταρχάς τι γνωρίζετε για τα όσα έκανε ο κυβερνήτης της Τράπεζας, ε, όχι μόνο όσον αφορά τη σημασία για τι ε, δραστηριότητε πελατών εκτό Ευρωζώνη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα, όχι μόνο για τον κίνδυνο νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, ε, ο οποίο ε, διαπιστώθηκε και από το δικαστήριο, αλλά και για την ίδια τη συμπεριφορά του κυβερνήτη τη Τράπεζα. ξέρουμε ότι προσφύγατε στο δικαστήριο και θέσατε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία στη Λετωνία. Αλλά το θέμα είναι πώ το βλέπετε εσεί και πώ φαντάζεστε ότι σε περίπτωση περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ε, για ε, παράνομη συμπεριφορά ενός κυβερνήτη κεντρικής τράπεζας ε, κράτους μέλους της Ευρωζώνης, ε, θεωρείται ότι θα μπορούσαμε να παρέμβουμε για να παυθεί από τα καθήκοντά του στα πλαίσια της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν γνωρίζει τα στοιχεία της έρευνας ε, για τη συμπεριφορά του κυβερνήτη Ρίψεβιτς. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα πρώτο σχόλιο. Άλλο η προστασία της προσωπικής ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όσον αφορά αυτή την πρώτη απέτηση συμμορφωθήκαμε με το άρθρο 14,2 14.2 που προβλέπει ότι οι κυβερνήτες των εθνικών τραπεζών θα χαίρουν κάποιες προστασίες, Δηλαδή ότι θα μπορούν να απαυθούν από τα καθήκοντά τους εάν δεν ε, πληρούν τις προϋποθέσεις ε, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους ή αν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ε, παραβιάσεις και αποφάσισαν να παραπέμψουν την απόφαση ε, της πάυσης ε, του κυβερνήτη στο δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση. Επ' αυτή τη βάση, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7 Μαρτίου του 2018 να παραπέμψει για τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν ε, και την ε, πάυση του ως κυβερνήτη ε, στο δικαστήριο, διότι θεωρήθηκαν ότι είναι πάυση των καθηκόντων του και θεωρείται ότι το άρθρο 14.2 δεν ε, τηρείται σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει προσφυγή και δεν έχουμε στόχο εδώ να παρέμβουμε στην ποινική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη στη Λετωνία και αυτό διευκρινίστηκε σαφέστατα σε δύο επιστολές τις οποίες έστειλα στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας. Από εκεί και πέρα βέβαια η εθνική έρευνα συνεχίζεται και έκτοτε μετά που παραπέφθηκε το θέμα στο δικαστήριο υπήρξε δίωξη αν δεν κάνω λάθος και η διαδικασία συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ε, η υπόθεση αυτή ουσιαστικά έφερε στο φως ε, το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος γενικότερα και νομίζω ότι αυτό το είπα και στην προηγούμενη ακρόαση. Πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και των αρχών καταπολέμησης νομοποίησης παρανόμων εσόδων που προς το παρόν είναι ε, εθνικές αρχές μόνο και γενικότερα μεταξύ των αρχών αυτών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτή είναι η μόνη δράση που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το ε, επίπεδο και μόνο έτσι μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες υποθέσεις και να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Έχω και μισό λεπτό ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται ότι δεν είχατε καμία πληροφορία για τον κίνδυνο διαφθοράς ε, του λετωνού κυβερνήτη πριν την παρέμβαση των ΗΠΑ. Και το δεύτερο τμήμα της ερώτησής μου, στο οποίο δυστυχώς δεν απαντήσατε, είναι όταν έχετε την αίσθηση, όταν έχετε την υποψία ε, για περίπτωση διαφθοράς ενός κυβερνήτη κεντρικής τράπεζας, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα έπρεπε να κάνει. Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην σωστή συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των φορέων που λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να διαφυλάξουμε και την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης και για να είμαστε και άμαμπτοι ε, όσον αφορά τα δημόσια καθήκοντά μας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερος αυτό το οποίο συμβαίνει και γι' αυτό αποφασίσαμε να παραπέμψουμε στο Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο την υπόθεση για να δούμε τι ενδιάμεσα μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε για να υπάρξει συμμόρφωση με την κατάσταση. Αυτά γνωρίζουμε. Βασίσαμε ε, το τι κάναμε σε αυτά τα οποία γνωρίζαμε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρατε τίποτα πριν την πάυση του. Διακόπτει ο πρόεδρος, συγγνώμη, έληξε ο, ο χρόνος. Ο Μπέρντ Λούκε. Καλημέρα κύριε Ντράγκη. θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Ντράγκη, στην συνέντευξη τύπου της 14ης έκτου στην Ρήγα, μιλήσατε για τη σταδιακή κατάργηση... Μπορείτε να με ακούσετε? Τη σταδιακή κατάργηση του APP, όπως ε, είπατε επίσης ότι το APP είναι ένα σύνηθε εργαλείο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα παραμείνει. Αυτό σημαίνει ότι επιφυλάσσεστε ανα πάσα στιγμή όπου θεωρείτε ότι πληρούνται ορισμένε ε, περιστάσεις να επαναλάβετε τις καθαρές αγορές ε, αξιογράφων. Δεύτερο, ποιο είναι το βασικό κριτήριο για τέτοια επανάληψη. Ο ρυθμός του πληθωρισμού ήδη έχει αμφισβητηθεί, αλλά ρωτήθηκε και από τον κύριο Χέκμαρκ. Ο ενίο δείκτη τιμών καταναλωτού στην Ευρωζώνη υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, για παράδειγμα, η αξία της κατοίκησης. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να ληφθούν υπόψη και θα μείωναν τότε τον ρυθμό πληθωρισμού από ό,τι είναι πραγματικά. Ορισμένες χώρες μέλη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της ιδιοκατοίκησης. Θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει μια στρέβλωση στον υπολογισμό του ρυθμού του πληθωρισμού και επομένως θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κριτήριο αυτό για μέτρα ε, για το APP. Δεύτερο, τα πραγματικά, πραγματικά επιτόκια στην Ευρωζώνη διατηρούνται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Σχεδόν μάλιστα είναι αρνητικά. Όμως αποτελούν σημαντικό εργαλείο κατευθύνσεως επενδύσεων και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των επενδύσεων. Θεωρείται το γεγονό ότι τα πολύ χαμηλά πραγματικά επιτόκια μπορούν να οδηγήσουν και σε μη παραγωγικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Πρόεδρος Ντράγκη, σας ευχαριστώ. Πρώτα, θεωρούμε ότι η νομισματική πολιτική έως τώρα είναι πολύ αποτελεσματική και τα προγράμματα αγοράς αξιογράφων. Δεύτερο, η απάντηση στην ερώτηση σας είναι ναι. Το πρόγραμμα APP αποτέλεσε εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Βρίσκεται στην εργαλειοθήκη μας και εάν προκύψουν περιστάσεις που να αιτιολογούν τη χρήση του εργαλείου θα το χρησιμοποιήσουμε. Επί του παρόντος δεν βλέπουμε τέτοιες περιστάσεις που να απαιτούν την παράταση ή επιμήκυνση του προγράμματος APP πέραν από το χρονικό όριο που ανακοινώθηκε στην συνέντευξη τύπου. Τρίτο, είναι αλήθεια και δεν αμφισβητούμε τους δείκτες τιμών καταναλωτού που επεξεργάζονται τα στατιστικά γραφεία της Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε ένα, μια, ένα, ένα οριμονισμένο δίκτυ τιμών καταναλωτού και όπως είπατε σωστά, αυτό δεν περιλαμβάνει τη διακατοίκηση. Τα έχουμε συζητήσει από την αρχή τα πράγματα αυτά, από την αρχή της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτα-πρώτα το πρόβλημα είναι και χρόνου και υπάρχουν και αντικειμενικές δυσχέρειες για να υπάρξει δίκτυς ο οποίος να περιλαμβάνει το στοιχείο αυτό. Υπάρχουν μελέτες απεικονίσεις που έχουν γίνει και δεν δείχνουν μεγάλη διαφορά. Ή πάντως όχι τέτοια διαφορά που να μην δικαιολογεί τα ε, ε, εργαλεία νομισματικής πολιτικής που είσαμε ως τώρα. Τέλος, το γεγονός ότι μπορούν να δημιουργηθούν εταιρείε ζόμπι, αυτό το εξετάζουμε εδώ και μερικά χρόνια κιόλα, διότι πράγματι αποτελεί μια ένα ενδεχόμενο. Αλλά δεν έχουμε δει πολλά τέτοια πράγματα. Πώς θα μπορούσαμε να είχαμε τέτοια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, όπως έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια και το 2017 ακόμη, εάν αυτή η ανάπτυξη είχε δημιουργηθεί από μαζικό αριθμό μη παραγωγικών επιχειρήσεων. Δεύτερη παρατήρηση. Βλέπουμε αυξανόμενη μόχλευση. Όχι, το αντίθετο. το, η μόχλευση κατεβαίνει, διότι χρησιμοποιούν χρήματα για να ξεπληρώνουν τα χρέη. Τρίτο, παρατηρούμε αυτό που λένε οι τράπεζες evergreening, δηλαδή χρηματοδότηση χρηματοδότηση ε, που δεν, οφειλετών μάλλον, που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Όχι, τα NPL μειώνονται, τα non-performing loans μειώνονται. Ευχαριστώ Καλώ ήρθατε στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Δύο ερωτήσεις. Θα γνωρίζετε αυτά που έχει γράψει ο Hans Βέρνερ Zinn, κυρίως σε ένα βιβλίο που έγραφε ότι το επόμενο κράχ, η κράχ θα είναι το κράχ του Ντράγκη. Όταν εξετάζετε την, τον, τους ιταλικούς στόχους. Τώρα, ναι, καλά, μου έχει γίνει και μόνη ιδέα. Αλλά αν εξετάσετε τον ιταλικό στόχο, θα δείτε ότι το χρέος είναι 500 δισεκατομμύρια. Τι είδους κρίση είναι αυτή. Και δείχνει, είναι δεικτικό κάποιων προβλημάτων στο σύστημα. Δεύτερη ερώτηση θα είμαι ο εισηγητής για την επόμενη τήση έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και στη Φιλανδία λένε, αν μεταφραστεί στα αγγλικά, βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα περίπου ας πούμε. Από τη μια μεριά λοιπόν εσείς εποπτεύετε τις τράπεζες, αλλά είσαστε κατά κάποιο τρόπο ο λύκος στα πρόβατα ή η κατσίκα στον κήπο. Το βρίσκεται ότι αυτό είναι πρόβλημα ή να ζητήσω κατανομή εργασίας στην έκθεση που θα συντάξω. Ευχαριστώ πολύ. Ας, ρωτήσω, ας απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Να κάνετε αυτό που θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ ότι να γράψετε στην έκθεσή σας. Μπορώ να σας πω ότι τα παραδείγματα θεσμών όπου έχετε και νομισματική πολιτική και εποπτεία είναι πολλά και πολυάριθμα και σημαντικά. Ας αρχίσουμε από την ε, Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, αλλά και άλλες χώρες όπως η Τράπεζα τη Αγγλία και ούτω καθεξής. Δεν είναι δηλαδή άνευ προηγουμένου. Δεύτερο, ειλικρινώς, δεν έχουμε δει καμιά σύγκρουση συμφερόντων και είναι και πολύ δύσκολο να τα φανταστεί κανεί και ω αφηρημένε έννοιε. Αν έχετε μια νομισματική πολιτική η οποία παρακολουθεί την εντολή της, τη σταθερότητα των τιμών και έχετε και μια εποπτεία η οποία επίσης στηρεί την εντολή της, της νομιματικής σταθερότητας και οτιδήποτε είναι σχετικό, σε πλήρη ανεξαρτησία της ΜΕΝΑ από τις δε, δεν υπάρχει καμιά σύγκρουση συμφερόντων, δεν προσπαθεί ο ένας να επηρεάσει τον άλλο, δεν μειώνουμε, όπως είπε κάποιος πριν, δεν αυξάνουμε τα επιτόκια επειδή θεωρούμε ότι αυτό θα διορθώσει την ε, νομισματική σταθερότητα. Δεν είδαμε κινδύνους για την νομισματική σταθερότητα που να μπορεί να ε, διορθωθεί με αύξηση επιτοκίων. Μόνο επιτόπου είδαμε κινδύνους. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σα ερώτηση, το έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας σα δώσω πρώτα μια ε, απάντηση γενική οι liabilities στόχου 2 έχουν αυξηθεί και ο λόγος είναι ότι πολλές τράπεζες μη, μη χωρών πυρήνα αγοράζουν αξιόγραφα από θεσμούς που δεν έχουν έδρα στην ίδια τη χώρα. 50% των ιδρυμάτων που είναι εκτός ζώνης ευρώ και 80% των πολιτών αυτών των αξιογράφων έχουν την έδρα τους εκτός των χωρών αυτών όπου, αγοράζονται οι ε, κινητές αυτές αξίες. Αυτό που έχει σημασία δηλαδή για τους ισολογισμούς στόχου 2 είναι πού ρυθμίζονται αυτές οι ροές και πού σημειώνονται, σε ποιους ισολογισμούς μπαίνουν. Είναι αδιαμφισβήτητο δηλαδή ότι έχουν αυξηθεί οι ισολογισμοί από την αρχή της αγοράς κινητών αξιών και θα μειωθούν όταν θα πάψει να λειτουργεί το σύστημα αυτό. Υπάρχει και μια άλλη πιο συγκεκριμένη απάντηση για το τι βλέπουμε στην Ιταλία. Ο αριθμός που βλέπουμε στην Ιταλία είναι μεγάλος, σημαντικός, αλλά όχι άσχετος με την ιστορική εμπειρία. Και πάλι διόλου χωρίς προηγούμενο. Άρα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Thank you, Ernest Thank you, Mr. President. Um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα μια επιστολή από 15 NG, ΜΚΟ και ζήτησε από την ΕΚΤ να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά τη διαφάνεια, την χρηματοδοτική, όσον αφορά του κινδύνου και τη συνέπειε αλλαγή του κλίματο. Στην επιστολή αναφέρεται η σημασία τη διαφάνεια και τη αποκάλυψη όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο και καλωσορίζει το ρόλο του Συμβουλίου για τη Χρηματοστατική Σταθερότητα που βάζει την αλλαγή του κλίματος στο αιματολόγιο, δημιουργώντας μια ομάδα για τη οικονομική αποκάλυψη στοιχείων. Δοθέντος ότι η ΕΚΤ έχει πάνω από 440 δις αξιόγραφα του ιδιωτικού τομέα μέσω των προγραμμάτων εξαγορά αυτών των αξιογράφων, ποια είναι η δυνατότητα η ΕΚΤ σαν δημόσιο θεσμικό όργανο να δώσει το παράδειγμα και θελοντικά να εφαρμόσει τις συστάσεις της Task Force για τις αποκαλύψεις στοιχείων σχετικά με το κλίμα. Θα ξεκινήσετε κάτι τέτοιο, θα το προτείνετε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΚΤ. Δεύτερη ερώτηση. Σε πρόσφατη ομιλία που κάνει στη Φλωρεντία, κυρία Ντράγκη, ζητήσατε αποτελεσματική αντικυκλική υποστηρίξη του συνολική ζήτηση. Μπορείτε να το περιγράψετε, ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μέσου και ποια χαρακτηριστικά και μεγέθη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να, είναι, να έχει μακροοικονομικά νόημα αυτό το μέτρο. Απάντηση. Να ξεκινήσουμε το δεύτερο ερώτημα. Η παρουσία κάποιου οικονομικού δυναμικού με σταθεροποιητικές δυνατότητες είναι πολύ σημαντικό για να ολοκληρωθεί η νομισματική ένωση και να καταστεί ανθεκτικότερη, λιγότερο ευάλωτη. Επίσης, στην ίδια ομιλία που αναφέρατε, είπα ότι όσο πιο πολλά έχει επιμερισμού του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα, τόσο λιγότερο χρειάζεσαι δημόσιους πόρους για να χρηματοδοτήσεις ε, τη λειτουργία σταθεροποίησης. Παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι μια εύρυθμη νομισματική περιοχή, ζώνη, 75% του κινδύνου μοιράζεται από τις ιδιωτικές χρηματοστικές αγορές και 25% μοιράζεται μέσω της λειτουργίας του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, δηλαδή πολιτείες ή μέλη το, τμήματα των ΙΠΑ που έχουν ύφεση αυτομάτως πληρώνουν χαμηλότερους φόρους και υπάρχουν άλλοι αυτόματοι σταθεροποιητές όπως είναι το, το σύστημα ασφαλίσεως για την ανεργία. Στην Ευρώπη το ίδιο στοιχείο είναι 40% Ιδιωτικό επιμερισμός του κινδύνου από τις χρηματοπιστικές αγορές και τα υπόλοιπα διαμοιράζονται μέσω της λειτουργίας των ε, κυβερνητικών προπολογισμών. Κατά κάποια έννοια, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η Ένωση των Κεφαλαγορών και η Τραπεζική Ένωση, τόσο μικρότερο θα είναι το μέγεθος ε, του δημοσιονομικού δυναμικού που απαιτούμε για να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μέσω της χρήσης δημοσίων πόρων. Πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό σημείο να το θυμούμαστε στι συζητήσει. Και είναι ένα τμήμα αυτού που προανέφερα, ότι η μείωση του κινδύνου και επιμερισμό του κινδύνου πάνε χέρι με χέρι. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και όχι όπως συζητούσαμε επί Μακρόν, που θεωρούσαμε ότι είναι δύο αντίθετε αντίθετες δυνάμεις. Για την πρώτη ερώτηση, να σας πω ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική, του στόχους της Ένωσης, υποστηρίζει τα συμπεράσματα της Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα. Επίσης υποστηρίζουμε άμεσα και έμεσα το συνεχιζόμενο έργο που λαμβάνει χώρα σε διάφορα διεθνή βήματα και συμμετέχουμε στο δίκτυο για το πρασίνισμα του χρηματοστικού συστήματος που συναδρίζει κεντρικές τράπεζες, εποπτικούς φορείς που θέλουν να έχουν διάφορες πρακτικές εποπτείας και συνετής διαχείρισης για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικούς και κλιματολογικούς κινδύνους. Τώρα τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εταιριών και της αγοράς των αξιογράφων τους έχουν καθοριστεί σκόπιμα ευρέως, ούτως ώστε να μην γίνεται διάκριση κατά των πράσινων ομολόγων Έχετε υπόψη ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατευθύνονται βασικά από νομισματικές πολιτικές και πτυχές αυτών και πρέπει να συμμορφωθούμε με την εντολή που είναι η σταθερότητα των τιμών. Όμως, η νομισματική μας πολιτική σίγουρα συμπεριλαμβάνει και τα πράσινα ομόλογα. Αγοράσαμε πολλά πράσινα ομόλογα και αγοράζουμε πολλά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είναι από τους μεγαλύτερους εκδότες πρασίνων ομολόγων στον κόσμο. Λοιπόν, τι προσπαθούμε να κάνουμε στα συμπέρασμα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα όρια που έχουν τεθεί και που προσανατολίζουν την νομισματική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Ήθελα κι εγώ να θέσω κάποιες πιο γενικές ερωτήσεις. Σε συνέχεια κάποιων ε, πραγμάτων που είπε ο κ. Χόκμαρκ. Καταρχάς, το 2011, όταν η ευρωπαϊκή οικονομία ξεκίνησε δειλά-δειλά την ανάκαμψή της, προσπαθήσατε να αυξήσετε τα επιτόκια. Ε, μάλιστα και ο προκάτοχός σας ε, προσπάθησε. Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί μια πολιτική η οποία περιορίζει την αύξηση των μισθών. Και κύριε Ντράγκη πρόσφατα ζητήσατε από τα συνδικάτα να είναι πιο απαιτητικά και να προσπαθήσουν να δουν αν μπορείτε να ε, ανακάμψει η κατάσταση, αλλά δεν ε, πέτυχε. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι η επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ παρά τα όσα γίνονται, έχει αφήσει ένα πληθωρισμό ο οποίος έχει σταματήσει σε επίπεδο το οποίο είναι χαμηλότερο από όσο θα έπρεπε. Και έχω τρεις άμεσες ερωτήσεις λοιπόν προς εσάς. Πρώτον, θεωρείτε ότι είναι λογικό να έχετε να αρχίσει να επαναχωρείτε σε κάποιες από τις πολιτικές, τις λίγες πολιτικές που έχουν αρχίσει να έχουν κάποια αποτελέσματα στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θεωρείτε ότι είναι σωστό να ζητήσετε απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Και τρίτον, σας ανησυχεί μήπως εκτραπεί η δημοσιονομική πολιτική λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και επίσης θα αυξήσετε τα επιτόκια ενώ σιγά σιγά θα αρχίσει να ε, σταματάει σταδιακά η ποσοτική χαλάρωση. Δεν πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί παραβίαση της ίδιας εντολής της ΕΚΤ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με το, τελε... Θα αρχίσω με το τελευταίο σας. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ζήτησα ποτέ <laughs> από τα συνδικάτα να ζητήσουν υψηλότερε αμοιβέ. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη των κοινωνικών εταίρων, όχι ασφαλώ των κεντρικών τραπεζιτών, να ζητήσουν ή να πούν στους κοινωνικούς εταίρου τι θα πρέπει να κάνουν ή να παραλείψουν. Όπως είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είμαστε πεπισμένοι ότι συγκλίνει ο πληθωρισμός και συγκλίνει και σε υπάρχει πλήθος προβολών, στατιστικών αναλύσεων, μελετών που το δείχνουν και συγκλίνει εις τρόπον που είναι και στη δηλαδή δεν χρειάζεται τη συνέχιση του Asset Purchase Program πέρα από τα χρονικά όρια που ανακοινώθηκαν στην ε, συνέντευξη τύπου για να μπορέσει να συγκλίνει ο πληθωρισμός. Και θεωρούμε ότι η πολιτική μας υπήρξε αποτελεσματική προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν από το τελευταίο Συμβούλιο ε, δείχνει καθαρά ότι θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και πέραν από την λήξη του ε, προγράμματος ε, αγοράς αξιογράφων και πέρα από το καλοκαίρι 2019, αλλά και παραπέραν χρειαστεί. Και το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να ρυθμίσει, να ε, ρυθμίσει τα ε, εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εισερχόμενα δεδομένα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πρόθεση, ούτε είπε κανεί τίποτε άλλο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια ή τίποτε σχετικό. Τώρα για τη δημοσιονομική πολιτική. Είναι σαφές ότι χώρες οι οποίες έχουν υψηλό χρέος θα πρέπει να έχουν βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική. Τώρα που η ανάπτυξη αρχίζει και τονώνεται, χώρες με υψηλό χρέος ιδίω θα πρέπει να ξαναφτιάξουν fiscal buffers, δημοσιονομικά περιθώρια δηλαδή, για την περίπτωση όπου η ανάπτυξη θα μειωθεί πάλι. Αυτή είναι και, αυτό μας διδάσκει η κρίση. Η κρίση έδωσε βέβαια πολλά διδάγματα. Ένα από τα οποία όμως ήταν αυτό. Οι χώρες οι οποίες είχαν ε, μεγάλο δημοσιονομικό περιθώριο, δηλαδή καλό δημοσιονομικό χώρο ήταν σε καλύτερη ε, θέση όταν τις έπληξε η κρίση. Δηλαδή μπόρεσαν να δαπανίσουν ας πούμε πολλά χρήματα για να ε, σώσουν τις τραπεζές τους. Άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο δημοσιονομικό περιθώριο και είχαν τραπεζικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν αργότερα δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο διότι οι αγορές πιστεύουν ή πίστευαν ότι η δημοσιονομική θέση των χωρών αυτών δεν ήταν βιώσιμη. η δημοσιονομικη θεση των χωρων αυτων δεν ηταν βιωσιμη κρίση λοιπόν μας διδάσκει πολλά πράγματα, αλλά πάντως ένα πράγμα που μας λέει είναι ότι εν ώψη του μέλλοντος, όταν η καιρή είναι καλή, καλά είναι να φτιάξει κανείς δημοσιονομικό ε, ζώνες προστασίας, buffer, για να μπορέσει να ανακάμψει. Όταν λάβει ο ήλιος, τότε βγαίνει, φτιάχνεις τη στέγη του σπιτιού, όπως είπε κάποιος. Αυτή ήταν και η άποψη τώρα για τη δημοσιονομική πολιτική. Τώρα, για τους μισθούς. Γιατί είμαστε επεπισμένοι ότι ο πληθωρισμός συγκλίνει προς την κατεύθυνση των στόχων μας και γιατί λένε το ίδιο και οι προβολές που κάνουμε. Διότι με τις προσδοκίες πληθωρισμού που είναι στέρεα δεμένες στον στόχο μας και με την οικονομία η οποία συνεχίζει σε πορεία ενίσχυσης βλέπουμε τις αγορές εργασίας να ενισχύονται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ενεργεία μειώνεται και βλέπουμε τους ονομαστικούς μισθούς να αυξάνονται. Το τελευταίο, τα πιο πρόσφατα νούμερα των ονομαστικών αποζημιώσεων ανεργαζόμενο είναι της τάξης του 2% για την ζώνη ευρώ από 1,6% προηγουμένως. Βλέπουμε λοιπόν τέτοια σημάδια και είμαστε πεπισμένοι ότι χάρη στην νομισματική μας πολιτική ο ε, ρυθμός του πληθωρισμού θα συγκλίνει προς τον στόχο που έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ. Μάρκο Βάλι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Ντράγκη θα ήθελα να συνεχίσω από την τελευταία απάντηση που δώσατε στην κυρία Μαρτίας ε, για τα ποσοστά της, ε, του πληθωρισμού, τα οποία λέτε ότι δεν είναι αυτά τα οποία λαμβάνετε υπόψη για την νομισματική πολιτική, γιατί λαμβάνετε υπόψη ε, το στοιχείο Island αλλά βλέπουμε ακόμα και τιμέ καυσίμων, για παράδειγμα, οι οποίες αυξήθηκαν ε, κατά ένα σημαντικό ποσοστό το τελευταίο διάστημα και ε, ήδη πρώτη ανάγκη ε, τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός είναι περίπου στο 0,91% τα ποσοστά αύξησης. Ίσως και σε ένα εγγύης μέλλον λοιπόν η τιμή των καυσίμων και μετά αυτών των αγαθών θα πρέπει να πέσει. Αναπόφευκτα λοιπόν θα αλλάξει και ο πληθωρισμός. Επομένως ο στόχος της σταθερότητας και οι τιμές της ΕΚΤ θα είναι μακριά από αυτό το στόχο του 2%. Εάν λοιπόν ο πληθωρισμός πάει προς αυτή την κατάσταση, η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει την πολιτική της και να επιστρέψει σε επεκτατική πολιτική. Και μία ακόμα ερώτηση, μιας και μιλήσατε και για την ε, μείωση των ε, μη εξυπηρετούμενων διανύων, των NPL. Ε, αυτό πρέπει να γίνει με κάποια ταχύτητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ευαισθησία για να μην υπάρχει και κερδοσκοπία για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, σε μία προοπτική μείωση των κινδύνων, κατά την άποψή σα είναι απαραίτητο να στοχεύσουμε και λίγο περισσότερο την προσοχή μας σε ε, τίτλους που έχουν ε, κατά βάση εμπορικέ ε, τράπεζες της Βόρειας Ευρώπης. Έχουμε μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής ΕΚΟΝ που διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κυρίως σε γαλλικές και γερμανικές εμπορικές τράπεζες και κατά την άποψή μου τώρα που είμαστε σε πιο ήρεμη αγορά αυτοί οι τίτλοι έχουν πολύ σημαντικό τίμημα και θα μπορούσαν ίσως ε, να χάσουν την αξία τους εάν βρεθούν στις αγορές. Ε, καλό είναι λοιπόν που θα υπάρχει ένας δείκτης στα επόμενα stretch test, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όπως γίνεται και για τα μη εξυπηρετούμενα ε, δάνεια και για αυτούς τους τίτλους δευτέρου και τρίτου επίπεδου. Θέλω να ξέρετε και την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. στην εισαγωγή μου, θα σας το ξαναδιαβάσω το κομμάτι που αφορά την ερώτησή σας και απαντά στην ερώτησή σας. Όταν αναφέρομαι στη μείωση κινδύνου και στον επιμερισμό κινδύνου, λέω ότι ο πρώτος ουσιαστικός ε, παράγοντας μείωση τη έχουμε ε, ένα βασικό στόχο των, ε, της υγείας των τραπεζών, ο οποίος είναι 67% υψηλότερος από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Περαιτέρω μείωση κινδύνου είναι καθοδόν, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των τοξικών ε, στοιχείων ενεργητικού στα χαρτοφυλάκια κάποιων μεγάλων ε, τραπεζών. Η απάντησή μου λοιπόν σε αυτό που είπατε είναι ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που μας είπατε. Όσον αφορά το ποσοστό του πληθωρισμού, το δεύτερο ερώτημά σας. Στις μελλοντικέ προβλέψεις προβλέπουμε μείωση των τιμών του πετρελαίου σε τέτοιο βαθμό δε που αναμένεται ότι ο πληθωρισμό για του επόμενου μήνε να βρίσκεται περίπου στο 1,5% και όχι στο 2% που είναι σήμερα. Αλλά ε, ο υφέρπον δείκτης ε, πληθωρισμού θα συνεχίσει να αυξάνεται και μάλιστα στις ε, προβολές που κάναμε για την τριετία βλέπουμε μείωση στις τιμές του πρεκρελίου αλλά αύξηση του υφέρποντος πληθωρισμού. Έτσι, ε, στα τέλη του 2020 ο πληθωρισμός αυτός θα είναι, ο συνολικός πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος και αν δεν κάνω λάθος θα είναι στο 2% ή στο 1,9% και ο βασικός πληθωρισμός Θα είναι ο πληθωρισμός δηλαδή, ο οποίος θα αποκλείει την ενέργεια και τα τρόφιμα. Αυτός είναι ο υφέρπον πληθωρισμός και έχετε και τον βασικό πληθωρισμό, ο οποίος θα είναι χαμηλότερος. Θα είναι 1,7% ή 1,8% στο τελευταίο τρίμηνο του 2020. Επομένως καλύπτεται αυτό που μας είπατε. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ σαφέστατος ορισμός. Υπήρχαν ε, διάφορες αποχρώσεις από ό,τι μάλλον συνομιτή. Γκέρολφ Άνεμανς. Όχι. Μπάρμπαρα Κάπελ. Δεν είμαι ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε Ντράγκη. Είπατε κάτι ενδιαφέρον σήμερα, ότι παρόλη την σταδιακή λήξη του Asset Purchase Program, θα συνεχίσετε την επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας παρακαλώ μας εξηγήσετε τι θα πρέπει να αντιληφθούμε. Δηλαδή, το ποσό του ισολογισμού που έχει φτάσει τώρα 586 δισεκατομμύρια θα ε, διατηρηθεί ή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Και έχω και μια άλλη ερώτηση για το, ε, ε, την, ε, την αντιμετώπιση εσωτερικού κινδύνου. Μιλούμε για το 41% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αναγκαίο know-how και τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσει και να φτιάξει σχετικά μοντέλα. Και σε ό,τι αφορά τις, α, τις τιμές ακινήτων, το APP είχε επιπτώσεις και στις τιμές που πληρώνουν ε, οι επιχειρήσεις για ακίνητα. Και ιδιωτικά και επαγγελματικά ακίνητα, ε, δήλωσε η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, είναι υπερτιμημένα κατά 35% μετά από τη λήξη του προγράμματος. Ποιες επιπτώσεις αναμένεται ιδίως στον τομέα των ακινήτων. Um, Επιτρέψτε μου να ξαναδιαβάσω αυτά που είχα πει όσον αφορά τα συμπεράσματα της πρόσφατης συνεντεύξεως τύπου. Αποφασίσαμε λοιπόν και προβλέψαμε ότι το Δικαιωτικό Συμβούλιο προβλέπει ότι μετά το Σεπτέμβριο θα μειώσουμε τις αγορές στοιχείων από 30 στα 15 δις και θα, τελειώσουμε το πρόγραμμα αυτό το Δεκέμβριο για την αγορά αξιογράφων. Και αυτό με την επιφύλαξη ε, άλλων στοιχείων που θα επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας για το μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Μετά αναφέρει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η νομισματική μας πολιτική θα γίνει λιγότερο επεκτατική διότι θα συνεχίσει να συνοδεύει την οικονομική ανάπτυξη επί χρονική περίοδο, γι' αυτό επιβεβαιώνουμε εκ νέου την επανεπινδυτική μας πολιτική. Ήτι τα χρεόγραφα που οριμάζουν θα ξαναγοράζονται για παρατεταμένη χρονική περίοδο και αυξήσαμε και τις καθεύθυνες γραμμές για τα επιτόκια. Είπαμε τα επιτόκια επί του παρόντος θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Ούτω Ούτως αποφασίσαμε. Περιμένουμε το και τη ΣΕΚΤ να παραμείνουν στο παρόν επίπεδο τουλάχιστον διαμέσου του θέρους του 2019 και εν πάση περιπτώσει το... τη χρονική περίοδο που απαραίτηται για να ευθυγραμμιστεί το ποσοστό του πληθωρισμού με τις τρέχουσες προσδοκίες για βιώσιμη διαδρομή προσαρμογής. Αυτή η νομισματική πολιτική ακροθυγός συνεζητήθη. Και αυτό το λέω να απαντήσει στην πρώτη μου ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση που ετέθη. Πόσο στενά παρακολουθούμε ενδεχόμενους κινδύνους. Μέχρι τώρα δεν βλέπουμε κάποια διολίστηση όσον αφορά τις κατηγορίες εξωγράφων. Κάποια όπως τα κίνητα, τα οι τιμές Τη στέγασης των σπιτιών, όπως είπατε, σε μεγάλες πόλεις, σε κάποιες χώρες και τα ομόλογα υψηλού απόδοσης και τα δάνεια μόχλευσης δείχνουν κάποιες διακυμάνσεις. Παρακολουθούμε αυτούς τους τομείς στενά. Ακόμα και η πρόσφατη διακύμανση, η υψηλή διακύμανση των χρηματοστατικών αγορών δεν επηρέασε αρνητικά όλα αυτά τα εξετάζουμε. Δεν νομίζουμε ότι δημιουργείται συστημικός κίνδυνος, αλλά τοπικοί κίνδυνοι που καλύπτονται και θα έπρεπε να καλυφθούν μέσω της μακρο μακροεργαλείων ε, συνετής διαχείρισης. Οι φυσαλίδες είναι πολύ ακριβές, έχουν συνέπειες μεγάλες όσον αφορά την οικονομία και όταν συνοδεύονται από υπερβολική ανάπτυξη των αύξηση των πιστώσεων. Όταν βλέπουμε αυτό, βλέπουμε ότι η αύξηση των δανείων, ε, η ανάπτυξη των δανείων ευθυγραμμίζεται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Εν γέννη λοιπόν, όπως ε, έλεγα στην αρχή της ακρόασης, δεν βλέπουμε να αυξάνεται η μόχλευση, η πίστοση, αυτό που χαρακτήριζε τα προηγούμενα έτη πριν από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Thank you, Gabriel Mato. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ως συνήθως κύριε Ντράκη είναι χαρά να σας έχουμε εδώ σήμερα. Να σας καλωσορίσω με τη νέα μου ιδιότητα ως εισηγητή για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, την οποία έχω ήδη αρχίσει να επεξεργάζομαι και θα ήθελα να προ... παρουσιάσω πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τρία θέματα θέλω να σχολιάσω. Καταρχάς ε, τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα ε, δάνεια. Είδαμε ότι είχαμε μία μείωση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ε, από το 8% πήγαμε στο 5,2% για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι στις χώρες μέλη, στις οποίες ε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας πλήττεται περισσότερο από αυτά τα κόκκινα δάνεια, δεν θα υπάρχει έλλειμμα ή μείωση της χρηματοδότησης, το οποίο θα οφείλεται ακριβώς ε, στα νέα μέτρα τα οποία καθορίζονται. Δεύτερο ερώτημα όσον αφορά την ε, προοδευτική απόσυρση των κινήτρων και την ανάγκη ε, να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το είπατε κι εσείς ε, και είδαμε ότι το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη έχει πέσει στο 8,4%. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η τάση, μια πολύ καλή τάση άλλωστε, θα μπορούσε να επισημοποιηθεί και να συνεχιστεί σε ένα σενάριο στο οποίο θα αποσυρθούν τα κίνητρα όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, κάτι το οποίο είναι από περιέργεια δική μου, τα κρυπτονομίσματα. Θεωρείτε εσείς, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα, ότι μακροπρόθεσμα η αγορά των κρυπτονομισμάτων θα, μπορέσει, θα συνεχίσει να αυξάνεται και μάλιστα να αποτελέσει και κίνδυνο για την νομισματική πολιτική και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δηλαδή, ε, σε τι ποσότητες ε, θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή κινδύνους ε, ε, και ποια είναι και τα ωφέλη αυτών των κρυπτονομισμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση όσον αφορά το κατά πόσον η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανέων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία. Είναι η ίδια ερώτηση που ετέθη πριν από κάποια χρόνια όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλοί ε, εποπτικοί φορεί ανά τον κόσμο πίεζαν τι τράπεζε να αυξήσουν ε, τα ποσοστά των κεφαλαίων του. Η απάντηση είναι αρνητική. Η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνει την κεφαλαϊκή κατάσταση των τραπεζών και σημαίνει ότι ο δανεισμό προς την πραγματική οικονομία θα είναι πιο επικερδής και θα αυξηθεί και μέσω πρόθεσμα. η προς την οικονομία. Και θα ήθελα να προσθέσω και το εξή. Για να μπορέσουν οι τράπεζες να ε, ε, συγκεντρώσουν κεφάλαια από τις ιδιωτικές αγορές, θα πρέπει να μειώσουν τα αποθέματα που έχουν σε κόκκινα δάνεια. Και μάλιστα αυτό που είδαμε και πρόσφατα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, είδαμε τράπεζες οι οποίες κατάφεραν να μειώσουν δραματικά τα αποθέματα που έχουν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μάλιστα κατάφεραν και με πολύ μεγάλη επιτυχία να αυξήσουν, ε, να συγκεντρώσουν ποσά κεφαλαίων από ιδιωτικά κονδύλια τα οποία θα ήταν αδιανόητα πριν από κάποια χρόνια. Υπ' αυτή την έννοια η μείωση λοιπόν των μη εξυπηρετούμενων δανείων συμπληρώνει ε, τη συνέχεια και την αύξηση του δανεισμού προς την οικονομία. Το δεύτερο φορά την απόσυρση των κινήτρων δεν αποσύρουμε κίνητρα στην ουσία. Η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι επεκτατική και το είπαμε και ότι χρειάζεται μεγάλος βαθμός ε, ε, νομισματικής ρύθμισης. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι αυτό θα συγκλίνει στο στόχο μας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει ε, το πρόγραμμα ε, αγοράς καθαρών στοιχείων ενεργητικών και την επιρροή του. Και το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε και μία αξιολόγηση και το διαπιστώσαμε αυτό και γιατί αυτό, διότι πιστεύουμε ότι η οικονομία είναι αρκετά ισχυρή για να συνεχίσει την επέκταση, παρά το γεγονός ότι το ΕΠΠ έχει μειωθεί σε σημασία μεν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ενισχύσει την ε, ε, καθοδήγηση για τα επιτόκια και συνεχίζουμε και τις επενδύσεις σε επαναγορά ε, ομολόγων τα οποία φτάνουν στη λήξη τους. Επομένως, ε, θέλουμε να συνεχίσουμε μέχρι το Δεκέμβριο το ΕΠΠ και την επενδυτική μας πολιτική για μεγάλο διάστημα και να συνεχίσουμε τα επιτόκια σε παρόν επίπεδο για τουλάχιστον, όπως σας είπα, μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Και από εκεί και πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να προσαρμόσει τα μέσα νομισματικής πολιτικής ανάλογα με το μεσοπρόθεσμο ε, ποσοστό του πληθωρισμού. Τέλος, για τα κρυπτονομίσματα. Καταρχάς, συμφωνούμε απολύτως ε, ε, με τις ανησυχίες της CSA, της άλλης εποπτικής αρχής, για την ανάγκη προστασίας των ε, επενδυτών και των καταναλωτών και μέτρα για τα κρυπτονομίσματα. Και τρίτον, κάτι που ρωτήθηκε προηγουμένως για την καταπολέμηση νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα μεγάλα ωφέλη των κρυπτονομισμάτων είναι ότι είναι ανώνυμα. Και επομένως πρέπει να υπάρχει δράση σε τρία μέτωπα. Βεβαίω δεν πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα αποτελούν κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα ποσά εξακολουθούν να είναι μικρά και η έκθεση των ε, ε, φορέων εποπτείας ε, στην Ευρωζώνη για τα κρυπτονομίσματα δεν έχει καμία σημασία, δεν, έχει, δεν θεωρείται ακόμα υπολογίσιμη. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διάδραση, διότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ένα αγαθό μέτρησης ή ένα καλό ε, μέσω πληρωμής, γιατί υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις και καταρχάς γιατί δεν υπάρχει κάποιο ε, χρηματοπιστωτικό όργανο το οποίο να ε, προστατεύει ε, τα κρυπτονομίσματα. υπάρχει η έκτη, η οποία προστατεύει το ευρώ. Ξέρετε ότι το ευρώ σήμερα θα είναι το ευρώ αύριο. δεν υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο για τα κρυπτονομίσματα, επομένως δεν μας ανησυχούν τόσο. Jakob von Weizsäcker. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ντράγκη. Ε, ερώτηση για το Nexus, για τον σύνδεσμο των, ε, ε, του δημόσιου χρέους. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Το καλό νέο είναι ότι θα έχουμε ένα fiscal backstop για το SAF. Εφόσον θα επιτρέψει, θα μάλλον θα, ε, αποτρέψει α, τους ε, ισολογισμούς να περάσουν. Αλλά βέβαια το κακό νέο είναι ότι ακόμα δεν έχουμε αντιμετωπίσει το αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή το δημόσιο χρέος να επηρεάζει το χρέος των τραπεζών, τις, ε, των των τραπεζών. Έχω ένα φάκελο, το NSBBS, και βασίζομαι στο SRB, τον SB, όπου θα δημιουργηθεί ένα fitness asset και με κανόνες για τους τραπεζικούς ισολογισμούς που θα επιτρέψουν να αντιμετωπιστεί το αντίστοιχο αυτό πρόβλημα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί προσεκτικά ώστε να μην προκαλέσει στρεβλώσει στι αγορές. Η ερώτησή μου είναι αυτή η στρατηγική πώς σα φαίνεται. Υπάρχουν και άλλες στρατηγικές βέβαια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όχι του sovereign nexus των τραπεζών, αλλά του sovereign nexus των τραπεζών. Thank you. Uh, well, first of all, we Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Τζάκη. Θα ε, πρώτα να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έχει κάνει. Θα ζητηθεί η γνώμη μας επ' αυτού και κατά τη γνώμη μου θα επανεξετάσουμε την πρόταση για τους τομείς που έχουν σχέση με την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί πλέον μεγάλη προτεραιότητα, δεν φαίνεται τουλάχιστον να είναι μεγάλη προτεραιότητα για τις χώρες μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκλίνει κατά κάποιους τρόπους από την έκθεση τη SRB High Level Task Force και ιδίως όλα τα SB tranches και τα junior θα αντιμετωπίζονται με ακριβώς ίδιο τρόπο σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα και για στόχους μεγάλης έκθεσης. Εν τέλει, αφενός δίνονται περισσότερα κίνητρα για την επένδυση σε αυτό το προϊόν, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί κινδύνους για, την, για τα non-senior tranches. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά ιδιωτική έκδοση των SBs. Εν τέλει, πρόκειται για μια καλή αφετηρία για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση η οποία φάνηκε ότι είναι παράγοντας αστάθειας όταν επέρχεται η κρίση είτε δημοσίου χρέους είτε τραπεζικού χρέους του συστήματος. Εν τέλει δηλαδή θα πρέπει να συνεχιστεί η εργασία στον τομέα αυτό και δεν νομίζω ότι έχουμε ακούσει και την τελευταία λέξη από αυτού. είναι κάπως ε, σαν δημοσιονομική ικανότητα, fiscal capacity. Και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ε, εργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Βάιτσεκερ, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει κανείς να εξετάσει το θέμα των αντοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν τα SPPS και ειδικά για το Junior Tranche. Έχω μεγάλη κατανόηση για την ε, γραμμή του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον θα ήταν να μάθω αν δέτε τα senior tranche, εάν αυτό είναι τρόπος οι ισολογισμοί του δημοσίου χρέους να μην υφίστανται μεγάλο κίνδυνο στην κατεύθυνση των τραπεζών. Και αν είναι ελκυστικός τρόπος αυτός για να προχωρήσει κανείς, κατά τη γνώμη σας. Σίγουρα το θέμα είναι κατά πόσο οι αγορές θα το ενστερνιστούν. Αυτή είναι η απαρχή του προβλήματος. Δηλαδή, να παράξουμε ένα αξιόγραφο το οποίο καλύπτει το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των κρατικών χρεών και που αγοράζεται επίσης από τις αγορές. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν τρόποι για καλύτερα senior transfers σε αυτό το βαθμό. Ευχαριστώ. Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Ντράγκη. Αγωνίζομαι εδώ και χρόνια για να υπάρξει ένας ορισμός του ρυθμού πληθωρισμού. Είπατε κάποτε ότι η μείωση των τιμών της ενέργειας προκαλούν αστάθεια. Λέτε τώρα ότι ο αριθμός πληθωρισμού είναι 2% χωρίς τις τιμές ενέργειας 1%. Οι τιμές της ενέργειας όμως συναποτελούν μέρος του πληθωρισμού και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μάθω με ποια μορφή σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ορίσει εκ νέου τον πληθωρισμό. Είτε κάτω του 2% για το σύνολο του πληθωρισμού, είτε ένα ασταθές μέρος και ένα βασικό πληθωρισμό, γιατί μέχρι τώρα αντιφατικά πράγματα έχω ακούσει, κατά τη γνώμη μου. Και επίσης, δεύτερο ερώτημα, προ δεκαετίας, μειώθηκαν, οι, ε, μειώθηκαν τα επιτόκια, πότε θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διότι μέχρι τώρα τηρούσαν ίδιο ρυθμό οι κεντρικές τράπεζες, ίδιο βήμα. ...769 εκατομμύρια στη Γερμανία... ...διότι εν τέλει αγόρασε η, ε, Γερμανική Κεντρική Τράπεζα ιταλικά ομόλογα. Ποιο όμω τώρα φέρει την ευθύνη για αυτά. Όσο υπάρχει το ευρώ και όσο δεν προκαλεί μεγάλα προβλήματα, μπορεί να πει κανεί ότι κάποια στιγμή θα εξισορροπηθεί. Όμω η τάση είναι σαφή. ώστε δικαιολογείται το ερώτημα πού βρίσκεται ο κίνδυνο και ποιο τον φέρει εν τέλει. Και τελευταία ερώτηση. Χωρισμός κράτους και τραπεζών. Αυτό το έχετε προπαγανδίσει εδώ και πολλά χρόνια. Χαμηλά επιτόκια όμως οδήγησαν στο ότι αυξήθηκε η κρατική συμμετοχή στις τράπεζες, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Γι' αυτό και η ερώτησή μου είναι εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε νέα όργανα όπως αυτά που εξήγησε ο κ. Βαϊτσέκερ, πώς θα ξεφύγετε από αυτήν την παγίδα. Πρόεδρος Δράκη. Σας ευχαριστώ. Ο στόχος μας είναι καθορισμένος σε ό,τι αφορά τον headline inflation, τον μετρούμενο πληθωρισμό, δηλαδή που περιλαμβάνει και την ενέργεια και την διατροφή, τα τρόφιμα. Εποτέ δεν υπήρξε σχετική αλλαγή. Παραπομπές σε, άλλα, σε άλλες μετρήσεις πληθωρισμού έχουν τη σημασία τους για να κατανοήσει κανείς πόσο σταθερή είναι η σύγκληση αυτή προς τον ρυθμό πληθωρισμού. Εξαρτάται από τιμές, γιατί μην λησμονείτε ότι η σύγκριση είναι μεσοπρόθεσμη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σταθερά. Εάν δηλαδή η επίτευξη του 2% πληθωρισμού οφείλεται σε ξαφνική αύξηση τιμών του πετρελαίου ή των τροφίμων και αναμένουμε οι τιμές αυτές να ξαναπέσουν, αυτό δεν σημαίνει ότι επιτυχάνουμε το στόχο μας διότι δεν είναι μεσοπρόθεσμη η αύξηση αυτή. Και εκεί μπορούν να παίξουν ρόλο άλλες μετρήσεις πληθωρισμού. Οι μετρήσεις πληθωρισμού που αποκλείουν τρόφιμα ή τιμές ενέργειας ή και άλλες, συλλαμβάνουν αυτό που συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, ανεξαρτήτως συστατικών των οποίων οι τιμές κυμαίνονται πολύ. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τις μετρήσεις αυτές για περαιτέρω πληροφόρηση για να μπορέσουμε να κρίνουμε σχετικά με την σταθερότητα της σύγκρισής μας. Εάν δηλαδή όντως είναι μεσοπρόθεσμη ή είναι μια έτσι μια αλλιώ. Touch and go. Εκεί συναντώνται οι διάφοροι ορισμοί, αλλά δεν υπάρχει σύγχυση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμά είναι ο μετρούμενος πληθωρισμός, headline inflation. Σε ό,τι αφορά τώρα τον στόχο 2, είπατε ότι είναι σαφής η τάση. Όχι, η τάση δεν είναι σαφής. Τώρα ανεβαίνει, ανέβηκε πριν, αλλά ξεκατέβηκε πάλι. Έχετε δίκιο στο εξή όμως. Οι χώρες οφείλουν να συγκλίνουν. Οι χώρες οφείλουν να προχωρήσουν σε διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρόκειται για ένωση η οποία βασίστηκε στο ότι θα έχει διαρκείς οφειλέτες και διαρκείς πίστοτες. Ο στόχος 2 λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά μέτρο των κεφαλαιοκών εκρόων. Είναι μέτρο που επηρεάζεται, όπως είπα και πριν, από το δικό μας πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Είδαμε να αυξάνονται ε, οι υποχρεώσεις. Θα δούμε την επόμενη ή τη μέθη επόμενη φορά σημαντική μείωση μέτρων στόχου 2, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μας πρόγραμμα αγοράς ε, ομολόγων. Και η τελευταία σας ερώτηση σχετικά με άλλα μέτρα ε, ας πω διαφορετικά η διασύνδεση μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζών φάνηκε ότι είναι παράγον που κατέστησε σοβαρότερη ακόμη την κρίση από ό,τι θα έπρεπε να ήταν. Μέτρα λοιπόν τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, είτε μέσω των ιδιωτικών αγορών για τα SB, είτε μέσω άλλων εποπτικών ε, μέτρων, θα είναι καλοδεχούμενα. Αλλά ας μην έχουμε ψευδεστήσεις, ότι δηλαδή αν έχετε μια σοβαρή κρίση δημοσίου χρέους, μια τράπεζα που δεν έχει καθόλου κρατικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό ό,τι είναι δίθεν ασφαλής. Αν έχετε μια σοβαρή κρίση δημοσίου χρέους, Όλοι θα πληγούν. Και οι τράπεζες είτε έχουν είτε δεν έχουν κρατικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους, αλλά και μη τράπεζες. Και ο λόγος είναι απλός. Όταν έχετε κρίση δημοσίου χρέους σημαντικού βαθμού, η ρευστότητα στερεύει. Το χρήμα φεύγει από τη χώρα. Οι τράπεζες χάνουν τη χρηματοδότηση. Είτε έχουν κρατικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκια του είτε όχι. Και το credit rating πέφτει δραματικά και εκείνη τη στιγμή όλα τα rating ακολουθούν το sovereign rating, την αξιολόγηση του δημοσίου χρέους. Επομένως, όλοι, τράπεζες, μη τράπεζες, οι παραγωγοί στην πραγματική οικονομία θα πληρώσουν πολύ περισσότερα για τη χρηματοδότησή τους. Όταν έχετε λοιπόν κρίση δημοσίου χρέους, αυτό πλήττει τους πάντες. Αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η Νίνα Τζίλ λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Καταρχάς, θέλω να μιλήσω για το Brexit. Τώρα που μιλάμε, η Στερλίνα πέφτει κάθετα, λόγω της παρέτησης του Υπουργού Εξωτερικών. Αλλά αφορά την αντιμετώπιση της αστάθειας. Με το Brexit και τη συνέχεια των συμβάσεων παραγόγων στην έκθεση δημοσιονομική σταθερότητα που δημοσιεύτηκε την περασμένη Τετάρτη, Τράπεζα τη Αγγλία είπε ότι η Βρετανική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί σε προσωρινό καθεστώ αδειοδότηση από το Μάρτιο 2019 και πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έκανε κάποια αντίστοιχη, δεν έδωσε αντίστοιχη υπόσχεση. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα για 29 3 παραγόγων, αξίες παραγόγων που δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας μετά το Μάρτιο του επόμενου χρόνου. Πρόεδρε Ντράγκη, Ποια είναι η απάντησή σας στην αξιολόγηση της Τράπεζας της Αγγλίας και την έκκληση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, επιβλέψει να επιτρέψει ένα καθεστώς προσωρινών αδειών. Δίκιο έχουν ή λάθος ότι δεν έχει προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Δεύτερον, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας στην επιστολή μας όσον αφορά τον αντίκτυπο του κλίματος στο πρόγραμμα αγορών του τομέα των εταιριών. Άκουσα σε πρώτερη απάντηση ότι πιστεύετε ότι το SPP έχει αγοράσει πράσινα ομόλογα. Πιο πέρα, θέλω για προς διευκρίνηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε μια ανάλυση του αντικτύπου που έχει το κλίμα όσον αφορά ε, το, την ποσοτική χαλάρωση, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και υπάρχει αξιολόγηση που έχει δρομολογηθεί από την ΕΚΤ διότι έγινε μελέτη του London School of Economics και λέει 62% από τον ομόλογα CFPP ε, βασίζονται σε ανθρακοβόρο τομέα κυρίως και σημαντικά. Μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πακέτο βιωσίμων χρηματοστητικών επενδύσεων. Το πακέτο όμως δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά επί κλιματολογικών στοιχείων και αποσιωπεί κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης. Εάν υπάρχει δυνατότητα συστημικών κινδύνων για μη βιώσιμες επενδύσεις λοιπόν, τι προτείνετε, πώς μπορούν όλα αυτά να εξομαλυνθούν. Απάντηση εκτός μικροφώνου του κ. Ντράγκη. Κάποιες από τις συμβάσεις που καθαρίζονται σε κεντρικό επίπεδο ίσως να έχουν πρόβλημα συνέχειας. Και διότι θα αλλάξει η νομοθεσία και θα αλλάξει τους ορισμούς των συμβάσεων και ίσως κάποια γεγονότα να επηρεάσουν τη ζωή των συμβάσεων στο μέλλον. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα, στις συμβάσεις που έχουν πρόβλημα. Αυτό εξαρτάται πόσα από, αυτά, από αυτές τις συμβάσεις θα εκπνεύσουν πριν από το Μάρτιο του 2019. Δεύτερον, εξαρτάται και από το αν κάποια πλευρά θα έχει νομοθεσία, η οποία νομοθεσία κατά κάποιο τρόπο θα μειώσει το πρόβλημα. Τώρα εδώ εκφράζω τη δική μας πλευρά, τις απόψεις μας. Εξαρτάται αυτό κατά πολύ από τι θα κάνουν οι ιδιωτικοί φορείς για να μειώσουν το πρόβλημα. Δεύτερον, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια ανάλυση του αντιχτύπου του προγράμματός μας ή πτυχών αλλαγής του κλίματος εντός του προγράμματός μας. Μπορώ να πω ότι θα το εξετάσουμε και θα δούμε ποια θα είναι συνέπεια. Ποια ήταν η τρίτη ερώτηση. Πώς οι βιώσιμες επενδύσεις μπαίνουν πιο πολύ στο, στο, βασικό τομέα επενδύσεων, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται περισσότερο επί των κλιματολογικών πτυχών και όχι επί των κοινωνικών πτυχών και των πτυχών ε, διακυβέρνησης. Απάντηση. Καταρχάς, καλωσορίζουμε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού. Καλωσορίζουμε και άλλες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Συμφωνούμε με την προτινόμενη ταξινόμηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στόχους της προτάσεως για τη βελτίωση της δυνατότητας αποκαλύψεως στοιχείων και βιωσιμότητα αυτών και να δημιουργηθεί νέα κατηγορία θε... Ε, βαθμολογήσεως με χαμηλή εκπομπή άνθρακα και με θετική εκπομπή στον αφορά άνθρακα, θετική βαθμολόγηση, αύξηση διαφάνειας και καλύτερη συγκρισιμότητα, αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε βιωσιμότητα και στη λήψη σωστών οικονομικών αποφάσεων, αποφεύγοντας μία απαραίτητη διαστρωμάτωση και επιβάρηση των χρηματοπιστωτικών κανονισμών και των νομικών κανονισμών. Συμφωνούμε και πολύ μάλιστα με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γιώργος Κύρτσος. Ε, πρόεδρε Τράγκη, Πρόεδρε Τράγκη, μετά το τέλος του ελληνικού προγράμματος έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι θέμα ε, και τι, τι μηνύματα θα στείλει. Επομένως, έχω τις εξής ερωτήσεις. Πότε εκτιμάτε ότι θα μάθουμε ή θα ολοκληρώσετε τη μελέτη της Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για το ελληνικό χρέος, την προοπτική του, την αξιολόγησή του. Η δεύτερη ερώτηση, και αυτή μεγάλου ελληνικού ενδιαφέροντος, είναι αν υπάρχει δυνατότητα, έστω σε μια καθυστερημένη, θα έλεγα, συμμετοχή των ελληνικών τίτλων στο QE, στο Quantitative Easing, το πρόγραμμα. Και το τρίτο, που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ την Ελλάδα και μας το, έθεσε, το θέσαμε μάλλον και στον κύριο Στουρνάρα σε πρόσφατη επίσκεψη ευρωβουλευτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, τι θα γίνει με το waiver, ε, αν θα παραμείνει δηλαδή, τώρα που η Ελλάδα είναι εκτός προγράμματος και από ό,τι μας είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, θα σας κάνει μια θετική εισήγηση, τέλος θα υποστηρίξει μια θετική άποψη ποια, είναι η θέση της τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να απαντήσω στις δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί στην ουσία πρόκειται για μία. Η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση αν έχει το waiver. Μόνο αν υπάρχει λοιπόν το waiver μπορεί να συμμετέχει. Τώρα, τα παρόντα προγράμματα ενισχυμένης εποπτείας ε, δεν εγγυώνται ότι θα υπάρχει το waiver και αυτό το διευκρινίσαμε. Αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε και εδώ έρχομαι να απαντήσω την πρώτη σας ερώτηση. Θα γίνει η δική μας ανεξάρτητη αξιολόγηση για την βιωσιμότητα του χρέους, ε, Debt Sustainability Assessment και θα δούμε και ε, θέματα διαχείρισης κινδύνου εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αυτό το waiver, την απαλλαγή και η ερώτηση που έρχεται σε συνέχεια αυτών είναι μετά από τα όσα αποφασίστηκαν από το Eurogroup με τα διάφορα μέτρα. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση τώρα όσο είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα πριν κάνουμε τη δική μας την αξιολόγηση όσον αφορά το θέμα αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση των διαφόρων κοινοβουλίων, τα οποία πρέπει να εγκρίνουν τις αποφάσεις οι οποίες ε, λήφθησαν από το Eurogroup. Και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένουμε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του EFSF μόνο μετά από αυτό μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους και την αξιολόγηση κινδύνων στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ο Γιάκοπ Φωμβάιτσέκερ. Ευχαριστώ πολύ. από την απάντηση στην ερώτηση του Έλληνα συναδέλφου, φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πριν από το 2032 ε, θα κάνετε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Τέλος πάντων, να συνεχίσω από κάτι που είπατε στο Βέρνερ Λάγκε. για το γεγονός ότι υπάρχει αντίκτυπος για τις τράπεζες από τα προβλήματα ε, χρέους, παρά το γεγονός ότι είναι τελείως διαφοροποιημένο το χαρτοφυλάκιό τους ε, για το ε, δημόσιο χρέος. Για παράδειγμα, η κρίση χρέους της Καλιφόρνιας δεν οδήγησε στα αποτελέσματα αυτά για τις τράπεζες της Καλιφόρνιας εμπειρικά. Και εδώ τίθεται το εξή ερώτημα, και αυτή είναι και η πρώτη μου ερώτηση προ εσά. Μήπω θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση αυτών των περιπτώσεων και να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του, στο, του κινδύνου αναδιάρθρωσης ε, δημοσίου χρέου που μπορεί να αντιμετωπιστεί, ε, μια έννοια που λειτουργεί κιόλα αποτελεσματικά και τον ε, κίνδυνο ο οποίος είναι πιο θεμελιώδης και δεν συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση της Καλιφόρνιας. Και σε αυτό το πλαίσιο τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Σκεφτείτε ότι αναφέρονται στην ενίσχυση της ασφάλειας, ε, της ε, άμυνας, ε, την προστασία των προσφύγων και ακόμα και θέματα κοινωνικής προστασίας. Ίσως δηλαδή θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτό σε μια περίπτωση στην οποία πράγματι μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο με την Καλιφόρνια σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Και όσον αφορά την πτυχή της κοινωνικής προστασίας, θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα πώς βλέπετε εσείς την ε, επίδραση της σταθεροποίησης μιας σοβαρής επανασφάλισης της ανεργίας. Δηλαδή θα έχουμε ένα σύστημα εθνικής αυτασφάλισης, ε, να υπάρχει ένα αποθεματικό ας πούμε για μια δύσκολη μέρα και ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη και τα όλα στοιχεία και τι, ανάλυση, τι δείχνει η ανάλυση σας, αν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά ε, ουσιαστική δυνατότητα σταθεροποίησης. Θα απαντήσω πρώτα την τελευταία σας ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό για πληθώρα λόγων που δεν χρειάζεται να τις αναπτύξω τώρα. Υπάρχει ένα συνδυασμό σταθεροποίησης και ταυτόχρονα μια κοινωνική διάσταση και συμβατότητα με την νομισματική ένωση και ενίσχυση της ε, εργατικής κινητικότητας. Είναι θετικό δηλαδή από όλες τις πλευρές. Βεβαίως πρέπει να σχεδιαστεί καταλήλως, πρέπει να λάβει υπόψη του και ε, τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συστήματα, πρέπει να λάβει υπόψη διαφορε... στην αγορά εργασία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν το συζητήσαμε αυτό βέβαια στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη σας παρατήρηση. Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας ή το παράδειγμα του Τέξας στη διάρκεια της, των κρίσεων της δεκαετίας του 80, μας λέει πολλά και μας δείχνει και πώς μια καλά ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση και μια ένωση κεφαλαγορών μπορεί να είναι ένας πολύ ισχυρό τρόπος να αποφύγουμε την εξάπλωση της κρίσης από τον τραπεζικό τομέα ε, σε ένα τοπικό σημείο προς την υπόλοιπη οικονομία. Στη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια πτώση των τιμών του πετρελαίου και πολλές από τις τράπεζες ε, του Τέξας χρεοκόπησαν και αυτό φυσικά έπληξε την οικονομία διότι ε, στέγνωσαν τα ταμεία. 20-30 χρόνια αργότερα στο μεταξύ και αυτό φυσικά συνέβη διότι η νομοθεσία τότε δεν επέτρεπε ε, ουσιαστικά στις υπόλοιπες τράπεζες των ΗΠΑ να ε, αγοράσουν το χρέος των τραπεζών του Τέξας. Ε, βέβαια αυτό άλλαξε και είχαμε μια ανθυρή αγορά τραπεζικών συναλλαγών από πολιτεία σε πολιτεία. Και φυσικά τα πάντα εξαρτώνται και από την ικανότητα του τραπεζικού συστήματα να δώσει δανειοδότηση, πιστώσει στην οικονομία. Και αυτό σημαίνει ότι ο επιμερισμό των κινδύνων μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό πριν καν σκεφτούμε το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια για τον επιμερισμό. Όσον αφορά τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ δύο μορφών ε, αναδιάρθρωσης του χρέου, εγώ είμαι μάλλον επιφυλακτικός. Όταν μπαίνουμε σε αυτά τα νερά, τα πάντα επηρεάζονται από τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι ο καλύτερος κανόνας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε μια κρίση χρέους. Δημοσιονομική σταθερότητα κλπ. είναι ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη, όπως θα είχε πει και ο προκάτοχός μου. Ευχαριστώ. Και ούτω ή άλλω υπάρχει και ο Ομοσπονδιακό Προπολογισμό, ο οποίο είναι κατά τι υψηλότερο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ομόσπονδο κράτο. Αν ε, αυτά λοιπόν μπορούν να οδηγήσουν ε, ε, σε κάτι καλύτερο, συμφωνώ μαζί σου. Ο Φούλβιο Μαρτουσέλο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη Μου φαίνεται ότι το τέλος ε, της ποσοτικής χαλάρωσης έχει διαφορετικές συνέπειες για την κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωζώνης μάλλον. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι θα σημαίνει αυτό για την Ιταλία. Και δεύτερη ερώτηση. Από το θεματολόγιο της κυβέρνηση εξαφανίστηκε παντελώς ε, η όλη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και τη μείωση του χρέου. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είχαν οδηγήσει σε επανειλημμένες παρεμβάσεις της ΕΚΤ, ε, λόγω της ανησυχίας βεβαίως ε, για τα ε, λογιστικά της Ιταλίας. Πιστεύετε ότι στο επόμενο διάστημα η χώρα μας θα μπορούσε να ε, επανεξετάσει τα θέματα αυτά. Καταρχάς να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Όταν αποφασίσαμε αυτά τα οποία αποφασίστηκαν στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, Τα αποφασίσαμε λόγω της ε, εκτίμησής μας ότι θα έχουμε σύγκληση ε, και ανθεκτικότητα της διαδικασίας του πληθωρισμού και ήμασταν βέβαιοι ότι η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη. Πρέπει βεβαίως να έχουμε κατά νου ότι η εντολή μας είναι η σταθερότητα των τιμών. Δεν είναι και δεν ήταν ποτέ να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, τα κέρδη των τραπεζών και μάλιστα μας επέκριναν διότι ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια μας και ε, τα κέρδη των τραπεζών ε, θα πληγούν, ε, το οποίο δεν συνέβη. Μπορεί να συμβαίνει βραχυπρόθεσμα, αλλά όχι μακροπρόθεσμα ή γιατί για να ε, προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ασφαλισμένων για τον ίδιο λόγο, επειδή τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά και τελικά ούτως ή άλλως μια χαρά πηγαίνουν από ό,τι βλέπουμε, διότι ναι μεν ανέλυβαν, ανέβηκαν ε, το κόστος ε, των ευθυνών, ανέβηκαν και τα στοιχεία ενεργητικού λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Επομένως, η αποστολή μας, η εντολή μας δεν είναι να προστατεύουμε τον εθνικό προϋπολογισμό της κάθε χώρας. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βεβαίως είμαστε βέβαιοι ότι η οικονομία ενισχύεται και όπως είπα και προηγουμένως η μείωση, η σταδιακή μείωση του APP συμπληρώνεται και από άλλα μέτρα νομισματικής πολιτικής και επομένως ε, υπάρχει ευρύ φάσμα δυνατότητας προσαρμογής και το είδαμε παρεπιπτόντως και από τις αντιδράσεις των αγορών στις αποφάσεις μας ότι δεν συνέβη τίποτα το δραματικό. Για τη δεύτερη παρατήρηση νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε πριν κρίνουμε. η δοκιμή θα είναι τα γεγονότα. Προς τον παρόν έχουμε ακούσει λόγια, άλλαξαν όμως και πρέπει να δούμε ε, πράξεις πριν ε, εκφράσουμε άποψη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, Περβάς Περές. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Δεν θα επαναλάβω την πρώτη μου ερώτηση. Στην υπόθεση θέλω να αναφερθώ αυτή που εφήγει από την Ίνα Γκίλ και από τον συνάδελφο Ορτασούν. Συμφωνώ μαζί σας. Η νομισματική πολιτική δεν επιδιώκει άλλους στόχους παρά μόνο την νομισματική πολιτική. Κάτι που συμπεριλαμβάνεται και συνθήκες και οριοθετείται εκεί. Δεν αντικαθιστά στόχους δημόσιας πολιτικής. Ούτε στη βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε όσον αφορά την υποστήριξη τη οικονομική δραστηριότητα. Αλλά στην ορθή πρακτική υπάρχει και μία ιδέα. Ποια, ο τρόπος εποπτείας των επενδύσεων Υπάρχουν επενδύσεις λοιπόν που λαμβάνουν χώρα και δημιουργούνται έτσι θετικές καλές πρακτικές. Πώς μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν στη στρατηγική της ΕΚΤ το reporting και το monitoring όσον αφορά την υποστήριξη των βιωσίμων επενδύσεων να μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν θέλω να αλλάξουν οι στόχοι της νομισματικής ε, πολιτικής, αλλά τι γίνεται με το reporting και το monitoring. Απάντηση. Ξέρω πού έγκυται το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είμαστε διαφανείς. Αρκετά διαφανείς όσον αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα αγοράς ε, ομολόγων και μπορούμε να δώσουμε συνολικά ποσά για τα βιώσιμα ομόλογα αλλά όλοι οι υπεύθυνοι της αγοράς μας λένε να μην αποκαλύπτουμε ξεχωριστά αναλυτικά ποσά διότι η αποκάλυψη θα έθετε κάποιοι συμμετέχοντες των αγορών σε θέση τέτοια που θα έχουν ειδικά ωφέλη λόγω της γνώσης. Θα αποκομίσουν ωφέλη. Οπότε η επίτευξη των στόχων της εντολής μας παρεμποδίζεται με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις όσον αφορά την υποβολή στοιχείων ομαδοποιημένων, συνολικών στοιχείων. Ο Ντάριο Ροζάτη, το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη που είμαστε μαζί σήμερα το απόγευμα. Δύο ερωτήσει έχω. Η πρώτη. Ορισμός της σταθερότητας των τιμών. Η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τον ορισμό σταθερότητας τιμών για τον καθορισμό της, του πληθωρισμού. Να είναι κάτω από το 2% πληθωρισμός ή κοντά στο 2%. Είναι ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην νομισματική πολιτική. Όμως, για τους σκοπούς ονομαστικής συγκλήσεως, αξιολογώντας επιδόσεις χωρών που είναι υποψήφιες, για την Νομισματική Ένωση, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί διαφορετικό ορισμό σταθερότητας τιμών. Το μέσο όρο τριών χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Θέλω να εκφράσω μια αμφιβολία. Δεν μπορείτε να έχετε δύο διαφορετικές έννοιες που αποδίδεται στον ίδιο όρο, όρο των συνθήκων. Στη συνθήκη Μιλάμε για σταθερότητα τιμών. Τελεία και παύλα. Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά. Μπορείτε να εξηγήσετε σε ποιο βαθμό είναι λογικό να χρησιμοποιούμε ε, δύο διαφορετικούς ορισμούς για δύο διαφορετικούς σκοπούς. Δεύτερη ερώτηση. Οι νομισματικές ε, συναλλαγές. Δεν είπατε κάτι πάνω σε αυτό. Θέλω να επιβεβαιώσετε ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να ισχύει και η ΕΚΤ εάν προκύψει ανάγκη, είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τον λόγο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση είναι αδιαφυσβήτητα ναι. Υπάρχει, ανήκει στην εργαλειοθήκη μας. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι τα δύο πράγματα είναι διαφορετικά, αρκετά διαφορετικά. Κοντά στο 2%, κάτω από το 2% ο μεσοπρόθεσμος στόχος αφορά τον καθορισμό, τον στόχο του πληθωρισμού που συνάδει με την εντολή μας για σταθερότητα τιμών. Ο άλλος ορισμός είναι να αξιολογηθεί η σύγκληση ενδεχόμενων μελλοντικών μελών για την Ένωσή μας. Ο σκοπός των δύο ορισμών είναι διαφορετικός. Ο ένας σκοπός είναι αξιολόγηση σύγκλησης, ο άλλος σκοπός είναι η προσμέτρηση α, της επίτευξης του στόχου, του στόχου. Μπορώ να συνεχίσω, να, κάνω, να δευτερολογήσω. Θέλετε υποψήφιες χώρες μέλη που θέλουν να γίνουν μέλη, θέλουν να συγκλίνουν τον πληθωρισμό τους και να πλησιάσουν το ε, πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας νομισματική πολιτική, έχετε στόχο πληθωρισμός να είναι στο, κάτω από 2% αλλά κοντά στο 2%. Δεν μπορείτε να έχετε δύο διαφορετικά είδη βαθμολόγησης. Δεν μπορείτε να ζητάτε τις υποψήφιε χώρες να έχουν χαμηλότερο πληθυσμό για να μπουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει. Τους λέτε, η συνθήκη ζητά πληθωρισμό κοντά στο μέσο όρο τριών χωρών που έχουν το χαμηλότερο πληθωρισμό. Μπορεί να είναι 0,1 πληθωρισμός. Θέλουμε αυτές οι υποψήφιες χώρες να έχουν πληθωρισμό 0,1% ή θέλετε να έχουν πληθωρισμό κοντά στο 2 αλλά κάτω από το 2. Απάντηση. Όπως προανέφερα, οι δύο καταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Και αυτό που είπατε για τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο πληθωρισμό, αυτή η διάταξη συνετάχθη όταν ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος και είχαμε κινδύνους από τον υψηλό πληθωρισμό. Θέλει να είναι κανείς σίγουρος ότι χώρες οι οποίες είναι υποψήφια μέλη να έχουν ένα πληθωρισμό που θα συγκλίνει προς το στόχο, υποθέτοντας ότι είναι άνωθεν προερχόμενες οι χώρες. Περί αυτού πρόκειται. Η σκοπή είναι εντελώ διαφορετική μεταξύ των δύο. Στη μία περίπτωση ε, ε, βασιζόμαστε στη σύγκληση βάση νομισματικής πολιτικής, στην άλλη έχουμε σύγκληση βάση των πράξεων των χωρών αυτών που κάνουν στις ανεξάρτητες πολιτικές τους μέχρι ότου να γίνουν μέλη της Ένωσης. Ο κύριος Νότης Μαριάς. Κύριε Ντράγκη, κύριε Ντράγκη, ήθελα να σας ρωτήσω για την απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό πρόγραμμα. Διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, το τρίτο πρόγραμμα προέβλεπε μια δανειοδότηση 86 δισεκατομμυρίων ευρώ και πολύ σκληρά μνημονιακά μέτρα. Τελικά τα μέτρα παρέμειναν, έγιναν ακόμη πιο σκληρά, αλλά τελικά υπάρχει ένα υπόλοιπο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ερώτημα είναι, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος, όπως αναφέρατε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε βέβαια όχι εις βάρος των ίδιων των δανειοληπτών. Θυμόσαστε ότι υπήρχε μια πρόβλεψη στο τρίτο δανειακό πακέτο 25 δις ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Χρησιμοποιήθηκαν όμως μόνο 4,5 δις. Το ερώτημά μου είναι απλό. Από αυτά τα 24 δις που περίσσεψαν, συμφωνείτε ένα μέρος να πάει για τη δημιουργία ενός ταμείου σωτηρίας των δανειοληπτών, ενός ταμείου που θα διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια με τέτοιο τρόπο ούτω ώστε οι δανειολήπτες να μην χάσουν τα σπίτια τους. Μια και περίσσεψε αυτό το ποσό. Αυτή την ερώτηση σας την είχα κάνει και πριν 1,5 χρόνο. Τώρα έχουμε τα δεδομένα, αυξημένα κόκκινα δάνεια, κίνδυνοι για πληστηριασμούς, αλλά ταυτόχρονα έχουν περισσέψει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρίτο δανειακό πακέτο. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε για να στηρίξουν τους δανειολήπτες, για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να έχω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Um, first of all... Πρώτα, πρώτα, δεν γνωρίζω ακριβώς τα νούμερα στα οποία αναφέρεστε. Και δεύτερο, δεν είναι δική μας απόφαση. Είναι απόφαση της χώρας μέλους. Τρίτη παρατήρηση. Αν μπορώ να παραφράσω κάπως ε, γενικότερα την ερώτησή σας. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημόσια χρήματα για να αγοραστούν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και ίσως στην τιμή ώστε οι τράπεζες να μην έχουν ζημία και τα άλλα μέρη να προστατευτούν οι οφειλέτες. Δεν είναι δυνατόν λόγω του ότι αυτό θα είναι κρατική ενίσχυση και δεν μπόρεσε να γίνει και σε άλλες χώρες που προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εμποδίζουν αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Μαριάς στα αγγλικά. Ε, έχουμε, όπως ξέρετε, την απόφαση της Κομισιόν το Μάρτιο φέτος, που καθορίζει τους όρους για τη δημιουργία μιας κακής τράπεζας. Τους όρους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση και αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Έχουμε την εμπειρία της Ιταλίας. Ρωτώ λοιπόν, μήπως στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος μπορούσε να υπάρξει αυτή η χρήση κεφαλαίων από αυτά τα 24 δις που περίσσεψαν επειδή είναι ειδικό πρόγραμμα για τη διάσωση υποτίθεται της Ελλάδος και έτσι να έχουμε μια ρύθμιση θετική για τα κόκκινα δάνεια. Ευχαριστώ. Σας είπα, δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν τα χρήματα αυτά υπήρχαν, ακόμα και αν τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταρχήν, θα υπήρχαν προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν και όλες οι άλλες χώρε σχετικά με τη δημιουργία κακών τραπεζών που θα αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια όχι στην εσωτερική τους αξία αλλά σε τιμές που δεν θα είναι τιμές της αγοράς. Γιατί αυτό είναι ο μόνος, ο μοναδικός τρόπος για να επιτύχετε το στόχο που λέτε και δεν είναι δυνατόν λόγω κανόνων που νομίζω, νομίζω συνήθως έχουν σχέση με την κρατική ενίσχυση. Τώρα μία ερώτηση για την μία, μία ερώτηση για την ποσοτική χαλάρωση, λέει ο κ. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το QE υπάρχει η δυνατότητα επίσης να ενταχθούν και ομόλογα, και ομόλογα των ελληνικών εταιριών, που είναι κάτι διαφορετικό ως πρόγραμμα. Επομένως, το ερώτημά μου είναι πρώτον, υπό ποιε προϋποθέσεις ομόλογα ελληνικών εταιριών μπορούν να ενταχθούν στο QE και δεύτερον, επειδή θα υπάρξει και πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που θα τελειώσει τον Αύγουστο του 2019, αν η Ελλάδα μπορεί να μπει συνολικά στο QE μέχρι τότε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι απάντησα πριν στην ερώτηση για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα, είτε χρειάζεται ένα waiver, μια εξαίρεση, ή θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους και κάποιες άλλες πτυχές διαχειρίσεως κινδύνου. Η θετικη αξιολογηση της βιωσιμοτητα του χρεους και καποιες αλλες πτυχε διαχειρισεω κινδυνου η εξαιρεση το waiver, θα εκπνεύσει με αυτό το πρόγραμμα και οι παρούσε διευθετήσει μετά το πρόγραμμα δεν επιτρέπουν εξαίρεση, waiver. Η η αυξημένη α, εποπτεία για μας, για να κάνουμε την αξιολόγηση, πρέπει πρώτα να δούμε ποιες θα είναι οι κοινοβουλευτικές απαντήσεις από κάποια κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του EFSF και σε αυτή τη φάση μπορούμε να το επαναξετάσουμε αυτό στα πλαίσια της δικής μας αξιολόγησης του DSA. Ε, και πιθανότατα και τα δύο θα είναι θετικά, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Επικρατεί μια αισιοδοξία έχουμε την πεποίθηση ότι θα μια, θα εφαρμοστεί μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πολύ θετικό και χρήσιμο για την Ελλάδα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ντράγκη υπό την ιδιότητά του που ήρθε σαν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας δέχομαι υπό την ιδιότητά σας σαν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Είναι φορέας αυτός για την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοστικού συστήματος στην Ένωση. Ο κύριος Τράγκη υπ' αυτή την ιδιότητα εμφανίστηκε τελευταία φορά τις 20 Νοεμβρίου του 2017. Δημοσιεύει SRB σήμερα την ετήσια έκθεση ε, για το έτος που τελείωσε 31 Μαρτίου. Έχει και σημαντικά θέματα, τα μακροπροληπτικά μέτρα που λαμβάνονται στην Ένωση θα εξεταστούν, κυρίως όσον αφορά το αντικυκλικό περιθώριο, τα συστήματα μόχλευσης και επενδύσει σε ταμεία ρευστότητα και ο κανονισμός που δημιουργεί αυτό το φορέα υπόκειται σε αναθεώρηση τη διαχείριση του κινδύνου. Και έχουμε πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συζητηθεί αργότερα την εβδομάδα στην Επιτροπή μα. Και αυτή η Επιτροπή του Διαχειρήσεω του Συστημικού Κινδύνου επέτρεψε να παρακολουθήσουμε τη συζητήση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν χώρα το τέλο Ιουνίου. Λοιπόν, μετά θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν την παρουσίαση γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 6 παρατέταρτο της εργασίας μας. Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά για μένα να σας απευθυνθώ την ιδιότητά μου που είμαι πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου Διαχειρίσεω του Συστημικού Κινδύνου. Σήμερα το ESRB δημοσιεύει την 7η ετήσια έκθεση που καλύπτει την περίοδο μεταξύ Απριλίου, 1η Απριλίου 2017 και τα 21η Μαρτίου του 2018. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την αξιολόγηση του κινδύνου τη μελλοντική του ESRB και κάνει μια ανάλυση και συζητεί τις συνεισφορές του SRB στην μακροπροληπτική πολιτική Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επίσης παρακολουθεί τη συνέχεια που δόθηκε στη στάση του SRB Καλύψαν πολλά από τα σημεία που καλύπτουν στην ετήσια έκθεση κατά τη διάρκεια προτέρων συναντήσεών μας. Γι' αυτό στα σχόλιά μου σήμερα θα ήθελα να εστιαστώ επί δύο θεμάτων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας δώσω μία σύντομη ενημέρωση όσον αφορά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, όσον αφορά τη μακροπροληπτική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, κινούμενοι προς την μακροπροληπτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήθελα να τονίσω τα βασικά χαρακτηριστικά των πρόσφατων συστάσεων του ESRB που έχουν σαν στόχο να αντιμετωπιστεί το θέμα ε, της ρευστότητα και της μόχλευσης και των σχετικών κινδύνων στα επενδυτικά ταμεία. Όταν συναντηθήκαμε τον περασμένο Νοέμβριο, σημείωσα ότι τέσσερες αρχές μακροπροληπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και αρχέ τη Νορβηγία και τη Ισλανδία, αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν αυτό τον αντικυκλικό, το αντικυκλικό περιθώριο, το ε, μέτρο απορρόφησης κεφάλαιο και τότε ελήφθησαν αποφάσει για θετικό τέτοιο μέτρο προφύλαξη στη Λιθουανία, Δανία, ε, Γαλλία και Ιρλανδία πρόσφατα. Και τώρα έχουμε 10 μέλη του SRB που προσπάθησαν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του τραπεζικού του τομέα εφαρμόζοντα αυτό το απόθεμα που κυμαίνεται από 0,25% το 2%. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση να είναι το νέο κανονικό, το νέο κανονικό όριο, λαμβάνοντα υπόψη τα χαρακτηριστικά στοιχεία του χρηματοστικού συστήματο και των οικονομικών κύκλων που ποικίλουν από χώρα σε χώρα και οι διάφορε ανοχέ των αρχών και οι προτιμήσει των αρχών για τον κίνδυνο, περιμένουμε ότι ένα υποσύνολο των αρχών θα χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο οποτεδήποτε. Τώρα θα στραφώ προ ένα άλλο τομέα, ο οποίο παραδοσιακά ήταν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων, ε, δηλαδή τα ακίνητα. Ε, παρατηρούμε ότι οι εθνικέ αρχέ συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ δραστηριοποιημένε όσον αφορά ε, τα ακίνητα για κατοίκηση. Μεγάλη πλειοψηφία 100 μελών έχουν τουλάχιστον ένα μέτρο που έχει σαν στόχο τα ευάλωτα σημεία αυτού του τομέα. Πολλές χώρες συνδυάζουν μέσα για να αυξήσουν την αντοχή των δανειοδοτών με μέσα που έχουν σαν στόχο την εγγύηση ε, ή τους δανειστές. Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε μόλι τώρα αναλυτικά πορίσματα σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σχετικά ζητήματα που αφορούν τον εμπορικό τομέα των ακινήτων και θα δημοσιεύσει μια έκθεση επ' αυτού του επόμενου μήνε. Ελπίζω να σα ενημερώσω επ' αυτού στην επόμενη συνάντησή μα. Όσον αφορά το έργο μας, όσον αφορά τον τομέα του επενδυτικού ταμείου, θα πρέπει να θυμόσαστε ότι πριν από ένα χρόνο ανέφερα σε αυτή την Επιτροπή έναν αριθμό κινδύνων που θα μπορούσαν να απορρεύσουν από τον αυξανόμενο ρόλο των επενδυτικών ταμείων ε, στην χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Το ESRB εξέτασε του κινδύνου ρευστότητα και του κινδύνου που σχετίζονται με τη μόκλευση και θεώρησε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η κίνδυνη. Το Φεβρουάριο αυτού του έτου το ESRB εξέδωσε μία σύσταση ούτω ώστε να καλυφθούν Αυτέ οι ανησυχίε για χρηματοστατική σταθερότητα, η σύσταση απευθύνεται προ ε, δύο μέλη, θεσμού μέλη, ε, η SRB, την Ευρωπαϊκή Αρχή για του Τίτλου και τι Αγορέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το SRB θεωρεί ότι η ΕΣΜΑ πρέπει να παράσχει στι εποπτικέ αρχέ κατευθυντήριε γραμμέ για να εφαρμόσουν τα μακροπληκτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Όμω, το ρυθμιστικό πλαίσιο επίση θα πρέπει να διευρυνθεί και προς αυτό το σκοπό συστήνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κάποιες ε, νέες ε, νομοθετικές, να κάνει κάποιες νέες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Η πρώτη ανησυχία απορρέπει το γεγονό ότι τα διάφορα εργαλεία για τη ρευστότητα που διατίθεται στα επενδυτικά ταμεία ποικίλουν πολύ σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαχείριση των διαφόρων μέσων ρευστότητας όπως τα τέλη αποκατάστασης είναι σημαντικά διότι βοηθούν τους διαχειριστές να αποκαταστήσουν τις διάφορες πιέσεις ε, σε... όταν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Η SSRB δεν θέλει να επιβάλλει τη χρήση κάποιων μέσων στα επενδυτικά ταμεία, όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ίδια ομάδα των εργαλείων είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, το SRB σε μια ανάγκη να αυξηθεί διεξαχθεί η δοκιμή αντοχής ρευστότητα στα επενδυτικά ταμεία και να διαδοθεί αυτή η κουλτούρα. Για αυτόν τον σκοπό η ΕΣΜΑ θα πρέπει να αναπτύξει προσανατολισμού για το πώ διαχειριστέ των διαφόρων ταμείων πρέπει να διενεργήσουν αυτά τα τεστ αντοχής. Θα πρέπει να υπάρχει και ανοιχτή. Θα πρέπει επίσης οι επενδυτικά ταμεία που έχουν λιγότερη ρευστότητα να δείξουν στου επόπτε ότι η επενδυτική στρατηγική μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και όταν υπάρχει ένταση στι αγορέ. Τρίτον, γνωρίζουμε ότι ενώ οι υποπτικοί φορεί είχαν τη δυνατότητα να περιορίσουν τη χρήση τη μόχλευση από εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το εργαλείο. Είναι σημαντικό η έλλειψη προσανατολισμού στον αφορά το σχεδιασμό του ενορίου να μην δημιουργεί ε, μια, μια κλίση προ την αδράνεια. Το SRB πρότεινε στην ΕΣΜΑ να αναπτύξει σχετικού προσανατολισμού. Τέλο, βρήκαμε ότι η έλλειψη εναρμονισμένου πλαισίου υποβολή εκθέσεων στα κράτη-μέλη αποτελεί εμπόδιο για την εποπτεία των διαφόρων επιχειρήσεων για συλλογικές επενδύσεις σε κινητούς τίτλους ή UCITS. Το ESRB συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων σε, σύστημα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα αποστείλουμε τις συστάσεις αυτές, θέλουμε να εφαρμοστούν γρήγορα, θα υποστηρίξουμε τους φορείς να εκτελέσουν το καθήκον και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει τον ρόλο του στην νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, θα παρακολουθούμε τι εξελίξει όσον αφορά τον τομέα των επενδυτικών ταμείων και στον ευρύτερο πεζικό τομέα να δούμε ποιε τάσει είναι αυτέ οι οποίε πρέπει να κατευθύνουν τι δράσει μα όφα την πολιτική. δική τη διαδικασία αυτή, το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε την τρίτη εκδοχή ε, του Shadow Banking Monitor που θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι με τα χαρά δεχτήκαμε την κυρία Περβάνς Μπερές και τον κύριο Μπούρκατ Μπάλτ, μια αντιπροσωπή από την παρούσα επιτροπή, στην τελευταία συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου του ESRB. Ελπίζουμε ότι αυτό ο τρόπο δημοκρατικής λογοδοσίας θα είναι υποφελής για την κυρία Μπερές και τον κύριο Μπάλτς όσον αφορά την επισκόπηση του ιδρυτικού κανονισμού του ESRB. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι τώρα διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για τη λογοδοσία εδώ η οποία ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρη μας. Να δώσω τώρα τον λόγο ε, στους συνεισηγητές. Ο κύριος Μπάλτς καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, εισαγωγική σας τοποθέτηση. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω περισσότερο που επιτρέψατε στην συνάδελφό μου Περβάνου Σουμπερές και σε μένα να έρθουμε την Φραγκφούρτη την προηγούμενη Πέμπτη και να είμαστε παρόντες και παρούσα δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για μας πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία και βεβαίως ε, εκφράζουμε και τη μεγάλη μας ικανοποίηση που είστε παρόν σήμερα εδώ. Υγείστε για 8η φορά, για, για 8η χρονιά, με συγχωρείτε, ε, του ε, Συμβουλίου και βεβαίω υπό διπλή ιδιότητα και ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπό την ιδιότητά σα αυτή, ε, ασφαλώ έχετε καθημερινά να ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι ανταποκρίνεστε πολύ καλά στα διπλά αυτά καθήκοντα. Το Συμβούλιο βρίσκεται κάπως σε δευτερεύουσα θέση απέναντι στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα ο κανονισμός προσφέρει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να έλθει και περισσότερο στο προσκήνιο. Είδαμε και από τον νέο μηχανισμό σταθερότητας SSM ότι υπάρχουν δομές μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ε, χρήση και αυτό θα ενισχύσει την θέση του θεσμού και θα επιτρέψει και την εντονότερη παρουσία της στην δημοσιότητα. Είναι σωστό να σκεφτεί κανείς με ποιο τρόπο μπορεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση του κανονισμού SRB. Γι' αυτό και η ερώτηση που έχω σήμερα προς εσάς είναι πώς μπορεί να δοθεί περισσότερη ορατότητα στον SRB από ότι μέχρι τώρα πώς μπορεί να γίνει πιο γνωστή η εργασία του SRB, του Συμβουλίου δηλαδή, όχι μόνο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και απέναντι στις κεφαλαιαγορές και ιδίως βέβαια στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Μπέρες. Δεν θα επανέλθω στην ε, επίσκεψη που ε, κάναμε παροιμήν ε, μαζί με τον Burkhard Μπάλτς. Ως συνεισηγήτρια θεωρώ την επισκεψή αυτή πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας προσφέρατε και που θεωρώ ότι δεν θα παραμείνει η μοναδική. Θα ήθελα ωστόσο να σας υποβάλω ερώτηση σχετικά με δύο πτυχές. Αφενός στην εισαγωγική σας τοποθέτηση δεν μιλήσατε καθόλου για τη λέξη Brexit, το B-word. Από συστημική άποψη, οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και αν η είσοδο στον προβληματισμό δεν είναι αναγκαία νομισματικού χαρακτήρα, μπορούν να οδηγήσουν σε αναταράξεις και άλλες ε, δυσκολίες των αγορών που μπορούν να έχουν τελικώ και συστημικό χαρακτήρα. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Δεύτερο, σχετικά με την πτυχή που αναφέρατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, σχετικά με, με για τη ρευστότητα και τις επενδυτικές ε, εταιρείες, ως γνωρίζετε, διαπραγματευόμαστε νομοθεσία που έχει προτείνει ο σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους όρους ρύθμισης και εποπτείας αυτών των επενδυτικών εταιριών με ένα διακύβευμα που είναι να γνωρίζει κανείς κατά πόσον η νομοθεσία της Βασιλείας εφαρμόζεται και μέχρι πού στην μεταφορά της στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ΕΡΒΕ και σε ΕΡΕΡ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά, τα θεμελιώδη στοιχεία που κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να βρουν θέση στην νομοθεσία αυτή, έχοντας υπόψη τους κινδύνους ρευστότητας και αυτή την ε, κακή εικόνα που μπορεί να έχει ακόμα ο ε, τομέας αυτός στην ευρωπαϊκή αγορά. Well, on, ε, <clears throat> on για την πρώτη ερώτηση που έλαβα, εάν το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο έχει μεγαλύτερη προβολή, συγγνώμη, το ε, Συμβούλιο έχει μεγαλύτερη προβολή, δεν χρειάζεται να κάνουμε αξιολόγηση κινδύνων. Πρέπει απλώ να δούμε τι πρωτοβουλίε θα ήθελε να δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτέ οι πρωτοβουλίε θα εφαρμοστούν και μάλιστα ταχύτατα. Εάν, για παράδειγμα, ε, αφορά το θέμα περισσότερη έκθεση στι χρηματοπιστωτικέ αγορές, έχουμε πάρα πολλού διάβλου που θα μπορούσαμε να ναι. χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό φυσικά ε, υπάρχουν και συνέργειες με πολλά μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων. Εάν το θέμα λοιπόν είναι η προβολή, απλώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πιο απλή οδό. Δηλαδή να αναφέρουμε τη σειρά των πρωτοβουλειών για την, να απευθυνθούμε για παράδειγμα σε χρηματοπιστωτικές αγορές ή σε υπομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλα βήματα τα οποία καταρχήν ε, γίνονται και μάλιστα πολύ εύκολα. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν ε, ε, για τις προτινόμενες αλλαγές της διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Αν έχετε ρωτήσει από αυτόν όμως, πολύ ευχαριστώ να τα σχολιάσω και αυτά. Τώρα για το Brexit. να πω ότι εξαρτάται πάρα πολύ ε, το πώς από το πώς θα το διαχειριστούμε. Στο τελευταίο ε, Διοικητικό Συμβούλιο κάναμε μια πρώτη συζήτηση για το Brexit και ε, το προσεγγίσαμε πάρα πολύ προσεκτικά, διότι υπάρχουν άλλα ε, βήματα στα οποία συζητώνται όλα αυτά τα θέματα και σίγουρα δεν θέλουμε να παρέμβουμε στις διάφορες διαπραγματευτικές θέσεις. Η συζήτηση που έγινε σε εκείνη τη συνεδρίαση για μένα ήταν πάρα πολύ εκπαιδευτική, διότι έδειξε ότι μπορούμε να συζητήσουμε το Brexit χωρί να παρέμβουμε στα όσα κάνουν οι υπόλοιποι. Ε, μπορούμε λοιπόν να διαβλέψουμε τους κινδύνους και μάλιστα και κάπου ξεχωριστά όπως γνωρίζετε, διότι συστήθηκε και μια τεχνική ομάδα εργασίας με την Τράπεζα της Αγγλίας για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους του Brexit εάν ε, ακολουθήσουμε το σενάριο του σκληρού Brexit. Και έτσι θα προχωρήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά οι συζητήσεις για το Brexit θα είναι όλο ένα και πιο συχνές ε, στην Επιτροπή τους επόμενους μήνες. Τώρα ως προς την ουσία. Όπως σας είπα, εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό ε, από τον τρόπο διαχείρισης. Αν δούμε τον αντίκτυπο της πραγματικής οικονομίας ε, του Brexit, θα είναι πάρα πολύ περιορισμένος ή μάλλον να το πω πιο προσεκτικά, θα είναι προς, ε, ε, περιορισμένος συνολικά. Υπάρχουν κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σίγουρα θα πληγούν περισσότερο, αλλά συνολικά και βραχυπρόθεσμα θα είναι περιορισμένος. Δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή τις οικονομικές συνέπειες μιας διαδικασίας την οποία δεν θα διαχειριστούμε σωστά και νομίζω ότι εδώ δεν είμαστε κι εμείς διαπραγματευτικός εταίρος, επομένως είναι καθήκον όλων των πλευρών σε αυτή την περίπτωση να εξασφαλίσουν ότι η ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς θα προστατευτεί, ότι η πρώτη δήλωση των ηγετών όπου θα έχουμε όλες τις ελευθερίες θα γίνει σεβαστή και από εκεί και πέρα ε, η διαπραγμάτευση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει κινδύνους χρηματοπιστωτικές ε, σταθερότητας, η οποία εν τέλει θα είναι και εις βάρος όλων. Ε, βεβαίως, σίγουρα κάθε φορά που το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω στοιχεία για το Brexit, αλλά εμείς δεν είμαστε διαπραγματευτικός εταίρος. Με ρωτήσατε συστάσεις για τη ρευστότητα και τη μόχλευση για τα επενδυτικά ταμεία. Σίγουρα πιστεύουμε ότι ένα διαφοροποιημένο σύνολο μέτρων ρευστότητας θα βοηθήσουν να έχουμε ε, σωστή διαχείριση των πιέσεων όταν θα δημιουργήσει πρόβλημα η ρευστότητα. Και επιπλέον η υπερβολική ρευστότητα και ε, θα πρέπει να μετριάζεται και θα πρέπει να προλαμβάνεται και έτσι θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να έχουμε συνθήκες ε, πίεσης της αγοράς και τι θα γίνεται. Τα, τα stress test λοιπόν ρευστότητα είναι πολύ σημαντικά εδώ. Όσον αφορά τη μόχλευση, Η καθοδήγηση ε, θα πρέπει να γίνει ε, αντικείμενο αξιολόγησης, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τα ε, μέτρα αξιολόγησης και αν μπορούμε να έχουμε εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Ευχαριστώ. Ο Νότης Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην λειτουργία των ασφαλιστικών... Do you have the interpretation? Okay. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, διότι αυτά, όπως ε, όλοι γνωρίζετε, παίζουν σημαντικό ρόλο και στην συστημική ευστάθεια και φυσικά στη λειτουργία της οικονομίας. Και το ερώτημά μου είναι πάλι σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα, τα οποία υπέστησαν ε, πραγματικά καταστροφή με το PSI το οποίο έγινε, υπέστησαν ζημιά τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξή Πρώτον, επειδή περίσσεψαν αυτά τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το δανειακό πακέτο των 86 δις, μήπως θα μπορούσε ένα ποσό κοντά στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ να αξιοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων όπως έγινε και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά υγιής λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων και να μην μειωθούν οι συντάξεις από 1η Πρώτου 2019 όπως αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup. Και μια τελευταία ερώτηση. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι μετά το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της αυξημένης εποπτείας, θα μπορεί να αποφασίσει και να μην εφαρμόσει τη μείωση των συντάξεων από η Πρώτου 2019. Είναι αυτή η εκτίμησή σας και η ανάγνωση της απόφασης του Eurogroup. Μπορεί η κυβέρνηση δηλαδή παρότι στα προαπαιτούμενα υπάρχει δέσμευση ε, να μειώσει τις συντάξεις από 1η Πρώτου 2019 να μην προχωρήσει τη μείωση των συντάξεων. Ευχαριστώ. Τα μέλη παρακαλώ να παραμείνουν στο, στο, Συμβούλιο του ESRB. Mr. Chairman, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Φεβρουάριο του 2016 το ESRB πρότεινε ότι οι ρυθμιστικοί φορεί μπορούν να κάνουν δοκιμέ αντοχή για του ασφαλιστέ και δεξιωτικά ταμεία για το θέμα του άνθρακα και του κλίματο. Δεν συζητείται δημοσία για τι δοκιμέ αντοχή απάντησε σε ερωτήσει του Κοινοβούλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδεχόμενη και παραθέτω εδώ πέρα ότι οι δοκιμέ για τον άνθρακα μπορεί να είναι χρήσιμο στοιχείο για να αξιολογηθεί η ε, σταθερότητα των χρηματοδοτικών ε, θεσμών και του συστήματο. Λοιπόν, πέρασε πρόσφατα ε, με διακομματική υποστήριξη ζητά το Κοινοβούλιο να θεσπιστούν δοκιμές αντοχής για τον άνθρακα όπως προτείνει το ESRB το 2016 για τράπεζες και άλλα χρηματοστικούς διαμεσολαβητές για να καθοριστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τέτοιου είδους στοιχεία ενεργητικού. Δοθέντως ότι υπάρχει ανανεωμένος ενθουσιασμός για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της νέας ταξινόμησης. Ε, πώς το λαμβάνει αυτό η υπόψη της ΕΡΜΗ για να αναπτύξει ένα σύστημα για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες για να κάνουν ε, δοκιμές αντοχής για τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις πρώτες δύο ερωτήσεις, όπως σας είπα δεν είναι δική μας απόφαση και ξανά όπως συζητήσαμε και προηγουμένως αυτό που πραγματικά δυσκολεύει τη χρήση των δημοσίων πόρων για ανακεφαλαίωση των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών είναι η νομοθεσία περικρατικών ενισχύσεων. Είναι η νομοθεσία περικρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπα, δεν είναι δική μα απόφαση και δεν μπορούμε να πούμε πολλά επ' αυτού. Το ίδιο θα ίσχυε και για την άλλη ερώτηση που είχατε για τι περικοπέ των συντάξεων και το πρόγραμμα τη κυβερνήσεω δεν είμαστε σε αυτό το, στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Ανήκει στο πρόγραμμα και τη συμφωνία μεταξύ τη κυβερνήσεω των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δεύτερο σημείο, τη δεύτερη ερώτηση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ε, το ESRB ξεκίνησε, δημιούργησε μια ομάδα ε, να επεξεργαστεί περαιτέρω το θέμα και να αναπτύξει μεθοδολογία για ε, εξέταση διαφόρων ενδεχομένων κάτι που θα διευρύνει τις αναλυτικές μα δυνατότητες εξολόγηση κινδύνων από την αλλαγή του κλίματος. Με τα χαράς λέω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ESRB μαζί με το Εποπτικό Δίκτυο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται το πρασίνισμα του συστήματος. Αυτό το έργο έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος, μάλλον μέχρι τον επόμενο χρόνο, να μπορώ να σα πω περισσότερα από αυτό. Λέτε ότι θα υπάρξει πρόταση που θα υποβληθεί του χρόνου. Αυτό μου λέτε. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Ντραγκή. Πρέπει να δούμε αυτή η ομάδα, η θεματική, τι θα παραγάγει και μετά ε, θα μπορέσω να πω περισσότερα για κάποιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που σας λέω και ε, μου, λένε ότι, ότι μόλις τώρα ξεκίνησαν τις εργασίες, αυτή η ομάδα συνεδρίασε μία φορά και μόνο. Ευχαριστώ, Μπερνάρ μόνο έχει το λόγο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα του συστημικού κινδύνου, να μιλήσω για τον εμπορικό πόλεμο που ασκούν οι ΙΠΑ κατά των ευρωπαϊκών εταιριών και μονομερείς οικονομικές ε, αβάσιμες ποινές επιβάλλονται. Η Γαλλική Τράπεζα, η PNP Paribas, ε, πλήθηκε το Μάιο το, το, το, 2014 από 9 δισεκατομμύρια δολάρια που επέβαλαν οι ΗΠΑ από εξοεδαφική ε, εφαρμογή αποφάσεως, αυθαίρετη κίνηση. Μπορεί να παραχθεί ένα πάσα στιγμή για οποιαδήποτε συστημική τράπεζα της Ευρώπης που έχει λιγότερα κεφάλαια από την BNP Paribas. Λοιπόν, ακόμα δεν θα υπάρξει λοιπόν οι καταθέτες των διαφόρων στόχων του Αμερικανικού συστήματος ε, θα υποστούν προβλήματα. Ε, οπότε θα δημιουργείται τραπεζικό πανικό αν σημειωθούν τέτοια προβλήματα με σημαντικέ ε, αποσύσει κεφαλαίων στην Ευρωζώνη. Το Φεβρουάριο του 2018 είδαμε σε μερικέ ημέρε τι μέσω η Λετωνική Τράπεζα MBLV τι έπαθε. με πάμε σε εποπτεία του SSM από Αμερικανούς εξοράστηκε και οι ρωσικές ε, εταιρείε επηρεάστηκαν. Όπως η Ρούζαλ παράγει αλουμίνιο τον Απρίλιο τον περασμένο επλήγει. Λόγω αυτών των κυρώσεων αυθερέτων που υπάγουν η και οδηγήθηκε στη χρεοκοπία με συνέπειε τιμικέ οικονομικές αγορέ, οικονομικέ αγορέ και διεθνεί. Οι Αμερικανικέ αρχέ μονομερό αποφάσισαν να αμφισβητήσουν και τι κυρώσει κατά του Ιράν. Οι Ευρωπαϊκέ εταιρείε ε, περισσότερο ποτέ διατρέχουν ένα κίνδυνο να τιμωρηθούν από αδικήματα που δεν έχουν διαπράξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλύψει τι ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες και του πελάτε, δίνοντα άμεσα πληρωμέ προ την Ιρανική Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το μονομερές λοιπόν σενάριο δεν μπορεί να αναπαράγεται ε, Μιλάμε για κυρώσει των Αμερικανών ε, που θα επιβληθούν έναντι 50 εταιριών όπου η ING που συμμετέχει μαζί με την Gazprom στο Nord Stream 2. Η Nord Stream 2 ε, διακόπτει ο προέδρο. Ασχολείται με το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο, παρέχει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Κύριε Μονό, μιλήσατε για δύο λεπτά. Θυμόμαστε τον αντίκτυπο που έχει η τη της Enron και τη WorldCom όσον αφορά τι οικονομικέ αγορέ το 2002, την εποχή που ήσασταν πρόεδρος του Φόρουμ Σταθεροποίησης. Διακόπτει ο προέδρο, δεν θα έχουμε διερμηνία. Τελειώνει η συνεδρία. Η ερώτηση για τον Πρόεδρο. Ερωτήσει για τον κύριο Ντράγκη. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Και διακόπτει ο κύριος Ντράγκη. Σε αυτή τη φάση δεν το συζητήσαμε ακόμα αυτό. Είναι σαφώς ένα θέμα και αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό Κοιτάξτε. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα και η κατάσταση παράξει κινδύνους για την οικονομική σταθερότητα, το ESRB θα πρέπει να το συζητήσει. Τι να κάνει. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι ή να προληφθούν οι κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τον Μαρκ Κάρτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Ντράγκη. Ευχαριστώ για τα αρχικά σας σχόλια. Δράτω με τι ευκαιρίε να πω εξ αρχή ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο με την ανταπόκριση στον αφορά το πόρισμα του δημοσιολαβητή για την κακή διαχείριση του κ. Ταΐς, του μέλους των G30 και καλό να τεθεί τέρμα στην σύγκρουση συμφερόντων και να φύγει πριν ο διαμεσολαβητής παραπέμψει το θέμα στο Κοινοβούλιο. Ερώτηση. Υπό την ιδιότητά σας, σαν πρόεδρος του ESRB, εάν η αγορά κινήτων της Ιρλανδίας υποστεί κλειδονισμό, έχει δημιουργηθεί φυσαλίδα, αυξήθηκαν οι τιμές ακινήτων και τα νίκια και διώχνει τον κόσμο την αγορά του τομέα. Όταν το έθεσα πέρσι, είπατε ότι η λύση για αυτή τη φυσαλία την ελληνική, για μια τέτοια αγορά που δεν είναι συστημική, είναι να επιληθεί μέσω τοπικής πολιτικής και μέσω κοινωνικής στέγασης στην Ιρλανδία. Νέε προειδοποίησει έχουν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δούνου του ΟΣΑ επί δύο θεμάτων. Κίνδυνο 10.000 αναδεθρωμένων στεγαστικών δανείων δεν θα είναι βιώσιμα αν τα επιτόκια αυξηθούν. Δεύτερον, ο κίνδυνος για την οικονομική σταθερότητα δημιουργείται από την υπεθερμασμένη αγορά κινήτων που τροφοδοτείται από διάφορα ταμεία αξιογράφων ιδιωτική αγορά που προσπαθούν να αγοράσουν αυτόν τον τομέα και να τοποθετήσουν σε κίνητα. Και τροφοδοτείται η πυρκαγιά αυτή που δημιουργεί προβλήματα. Ερωτήσει. Ποια είναι η άποψή σα, ποιο θα είναι ο αντίκτυπο αλλαγή επιτοκίων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια στην Ιρλανδία. Έχετε συστάσεις. Για να μειωθεί η φυσαλίδα κανονικά στον τομέα των ακινήτων στην Ιρλανδία. Το ESRB θα δημοσιεύσει κάποια προειδοποίηση ή ε, τεκμηριωμένη γνώμη που απευθύνει προς την Ιρλανδία όσον αφορά τους δημιουργουμένους κινδύνους στην παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ, Μπαρμπαρα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και εσά, κύριε Πρόεδρε Ερώτηση για το Brexit. Γνωρίζουμε ότι από χθε ε, την συνάντηση Βρετανική Κυβερνήσεως στο Checkers ότι υπάρχει ένα σενάριο αποχώρησης όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα παραμείνουν μέσα στην έννοια αγορά. Μόνο οι ανταλλαγέ αγαθών αυτό το ειδικότερο σενάριο, δηλαδή όπου οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε θα βγουν εκτός ενίας αγορά, Ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι μπορεί να έχει το σενάριο αυτό στην νομισματική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Δεύτερο, μέγα θέμα, πολλά δισεκατομμύρια, το χρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Με αυτό το νέο σενάριο πάλι ποιε επιπτώσει μπορεί να έχει. Τρίτο, μετά την αποχώρηση, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Τράπεζα της Αγγλίας θα έχουν καθεστώς παρατηρητού στο SRB, στο Συμβούλιο δηλαδή Συστημικού Κινδύνου. Thank you. Πρόεδρος Δράγκη, σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας που αύξησε το κεφαλαιοκό buffer από 0 σε 1% την προηγούμενη εβδομάδα μόλις. Να λοιπόν μία πρώτη απάντηση σε αυτό που είπατε. Γενικότερα πάντως το ερώτημα αυτό τίθεται και σε άλλα πλαίσια όπου βλέπουμε ότι οι αξιολογήσεις στέγης είναι μεν ε, τοπικά σε ορισμένες μεγάλες πόλεις αστικά κέντρα ε, υπεραξιολογημένες. Το ίδιο ισχύει όμως και για τον ε, εμπορικό ακίνητο. Για το πρώτο, σύμφωνα με την ανάλυση του 2016, το Συμβούλιο είχε εκδώσει προειδοποίησεις προς 8 χώρες, οι οποίες έδειχναν υψηλή χρέωση για τη στέγη και υψηλό κόστος στέγης. Για το εμπορικό ακίνητο είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα και ευρύτερο ε, όσον αφορά ε, το φαινόμενο. Για το εμπορικό ακίνητο η τροτότητα έχει σχέση με την προσπάθεια των επενδυτών να επιτύχουν απόδοση. Επομένως οι τιμές έχουν αυξηθεί και σε ό,τι αφορά και ιστορικές συγκρίσεις και ιδίως στις πρωταρχικές αγορές και τις έχουν καταστήσει ευάλωτες στο repricing και σε απότομες αλλαγές στην ε, στα risk premium. Παρόλο που οι τράπεζες έχουν σημασία και οι μη τράπεζες και η διαμεθοριακή χρηματοδότηση αυξάνει το ρόλο της. Λόγω λοιπόν της αύξησης των σημασιών του, του μη τραπεζικού τομέα είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν θα πρέπει να διατεθούν νέα μακροπροληπτικά εργαλεία και για εκθέσεις μη τραπεζών σε, ε, στην ε, έγκυο ιδιοκτησία, στη στέγη στο ακίνητο γενικότερα. Μακροπροληπτικά λοιπόν εργαλεία για μη τράπεζες, διότι προσφέρουν τη δυνατότητα άσκηση δραστηριοτήτων που μοιάζει πολύ με τραπεζικέ. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και οι βασικοί χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές. Αυτά για την πρώτη σα ερώτηση. Για τη δεύτερη, να σα πω το εξή κάτι το οποίο έχω πει και άλλη φορά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να σχολιάσει κανείς κάποια ενδεχόμενα τα οποία έχουν μεν συζητηθεί αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη. Για να είμαστε πιο σαφείς, εάν αυτή η ακαιρεότητα της ενιαίας αγορά πρόκειται να διατηρηθεί, θα εξαρτάται αυτό από την τελική ρύθμιση. Κάποιες δραστηριότητες θα φέρουν διαβατήριο και κάποιες άλλες όχι. Και αυτό θα είναι μία από τις επιπτώσεις αυτής ε, της συναλλαγής. Όμως η τελική διαπραγματεύση ακόμη δεν έχει γίνει, ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε, να εκφράσουμε άποψη για κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, για το καθεστώς παρατηρητού της Τράπεζας Ακρίας δεν το έχουμε συζητήσει αυτό ακόμη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Μπάρτς. Σας ευχαριστώ. Σύντομη ερώτηση. υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες κεντρικών τραπεζών και πολλή ικανότητα, πολλή γνώση κεντρικών τραπεζών στο Συμβούλιο SRB. Υπάρχει σε αυτό και ο κίνδυνος, ωστόσο, να είναι κάπως μονόπλευρη η γνώση. Ερώτηση προς εσάς, κύριε Πρόεδρε. Εάν ίσως πρέπει να υπάρχει ευρύτερη τεχνογνωσία, πέραν δηλαδή από τους κεντρικούς τραπεζίτες, με συμμετοχή από τους χρηματοπιστωτικούς επόπτες, για παράδειγμα, στο μέλλον και αν αυτοί θα πρέπει να μπουν επίσης στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Ο Πολτάνκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Ντράγκη. Νομίζω ότι η έκθεση του 2016 είναι αρκετά καθυστερημένη και αρκετά δημοφιλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην έκθεση πρωτοβουλίας για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση και μάλιστα αναφέρεται και στις τροπολογίες ε, για το CRR και το CRD όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να συμπεριλάβει τους συστημικούς κινδύνους ε, των στοιχείων ενεργητικού στο προληπτικό πλαίσιο. Δεν φαίνεται όμως να σας αρέσει εσά ιδιαίτερως. Όποτε σας ακούω να απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις, φαίνεται να την ξεχνάτε. Και ποτέ δεν αναφέρεστε σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού που πιέζονται. Πιστεύετε λοιπόν ότι ε, ε η έκθεση αυτή που είναι πάρα πολύ καλή θα έπρεπε να προχωρήσει. Και πώς θέλετε εσείς να προχωρήσει από το ίδιο, την ίδια την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα αντιμετωπίσουμε την, το, περίπτωση αυτών των στοιχείων ενεργητικών. Η πρώτη ερώτηση. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στην ε, Επιτροπή είναι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι τρία ψήφοι από τα 37 μέλη. εσεί εμεί δεν λέμε στην Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου τι να κάνει. Τρει ψήφου έχουμε. Μετά έχουμε του τρει προέδρου τη ε, Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, τον πρόεδρο τη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και μετά τα τρία ESA. Κεντρικές τράπεζες λοιπόν, αλλά όχι μόνον. Απλώς ε, εξηγώ ότι έχουμε πληθώρα πραγμάτων. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σε εθνικό επίπεδο, 19 κράτη-μέλη έχουν ε, ορίσει τις κεντρικές τράπεζες ως την αρμόδια αρχή για τη μακροπροληπτική προλητική ε, στον τραπεζικό τομέα. Εάν λοιπόν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και πούμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε και στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, ε, περισσότερο από άλλες αρχές. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν η σύνθεση της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου είναι αρκετά ικανοποιητική. Ε, η άλλη απάντηση είναι ότι δεν ήξερα ότι ε, εγώ ε, διστάζω να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι Εδώ τώρα απαντάω μόνο ως Επιτροπή Συστημικού Κιδίνου, Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετίζεται και από δουλειά που έχει κάνει η Επιστημονική Επιτροπή, ε, η Συμβουλευτική της Επιτροπής μας και όπως είπα και προηγουμένως έχουμε συστήσει μια ομάδα για να εξετάσει πιθανές μεθόδους ε, ανάλυσης των σενάριων και επομένω υπάρχει αυτή η ομάδα εργασία. θα εξετάσει τι διάφορε εκδοχέ και τι διάφορε μεθοδολογίε, θα δούμε τι θα προκύψει, αλλά εάν εσεί έχετε κάποιε άλλε προτάσει για το πώ θα μπορούσε ένας, μια επιτροπή, σαν την επιτροπή συστημικού κινδύνου που εξετάζει μακροπροληπτικά εργαλεία και έχει όλε αυτέ τι αρχέ γύρω από το τραπέζι, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, Εμεί είμαστε διατεθειμένοι. Ε, ο κύριο Τάνκ, η έκθεση λέει ότι ε, δεν θα πρέπει να έχετε μόνο μεθοδολογία για τα stress test, αλλά και τα εργαλεία για να περιορίσετε τον κίνδυνο, τον κίνδυνο παραδείγματος χάρη κεφαλαίκες απαιτήσει ή ε, όρια έκθεση. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί να τα συμπεριλάβει στο CRD και δεν βλέπω ούτε την Επιτροπή ή κάποιον άλλο να κινείται προ την ίδια κατεύθυνση. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Συστημική Κινδύνου δεν έχει ισχύ να επιβάλλει πράγματα. Ω αποτέλεσμα λοιπόν ε, τη Task Force και του τι θα κάνει, μπορεί να κάνουμε κάποιες προτάσεις για τα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά ε, πρέπει να πάνε όλα αυτά σταδιακά. Πρώτα θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα και μετά να προτείνουμε τα εργαλεία ε, ίσως θα μπορούσατε να πείτε και ότι ορισμένες φορές προχωράμε πάρα πολύ αργά. Ε, είναι και η δουλειά σας. Οι νομοθέτες κινούνται πάρα πολύ αργά. Είναι τμήμα της δουλειά σας ως πρόεδρος της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Ε, δείξτε και λίγη ανυπομονησία, δεν πειράζει. εντάξει, το σημειώνω, λέει ο κύριος Ντράγκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη για τα πολύ ε, θετικά στοιχεία που είχαμε στην ανταλλαγή απόψεων με τις δύο ιδιότητές του. Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση ε, την Τετάρτη 9 ώρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ.